à euh, euh, un groupe commun avec euh, Hans-Jörg Haber, qui est habitué de notre sous-commission, qui dirige la CPCC. Monsieur Lopez Blanc. Καλημέρα σας. Σας παρουσιάζω τον κύριο Τεκερκόβ, ο οποίο είναι υπεύθυνο για τα θέματα εξωτερικών υποθέσεων και τον κύριο Τεκερκόφ, ο οποίο είναι υπεύθυνο για τα θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στην περιοχή του Σαχέλ δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις νέες αποστολές οι οποίες έχουν ήδη εκκινήσει όπως ε, ισχύει για τον Ήγερα ή αυτές οι οποίες θα προβλέπετε, προβλέπετε να λειτουργήσουν όπως το Μαλί που είναι ε, αποστολές υποστήριξης σε θέματα ασφάλειας. Πρόκειται για αποστολές οι οποίες έχουμε επιζητήσει εμείς εδώ και πολύ καιρό, ίσως υπερβολικά πολύ καιρό, γιατί ίσως έχουμε επιμείνει περισσότερο στην διάσταση ασφάλειας των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πολι... έναντι των χωρών του Σαχέλ, κάτι το οποίο άργησε να ληφθεί υπόψη από τα κράτη-μέλη. Το σχέδιο ήταν γνωστό. Οι απειλές επίσης ήταν γνωστές. Με τον κύριο Ντεκερκόφ είχαμε συζητήσει για τα θέματα αυτά. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Από την στιγμή που από το Μάρτιο του 2011 υπήρχε στρατηγική για το Σαχέλ στο τραπέζι του Συμβουλίου, έχει περάσει ένα μισή χρόνο μέχρι το Δεκέμβριο σχεδόν του 2012 για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική. Είναι μακρύ αυτό ο χρόνο. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μα για την εκκίνηση αυτή τη αποστολή. Δεν έχουμε βέβαια μαγικά ραβδάκια για να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Είναι πολύ εύθραυστη και ασταθής η κατάσταση. Η διαδικασία του ΟΗΕ σε πολιτικό επίπεδο η οποία συνεχίζεται γιατί έχουμε το ψήφισμα 271 υπό το κεφάλαιο 7 της χάρτας του ΟΗΕ και ζητά από τις αρχές ε, του Μαλή να υποστηρίζει τις αρχές του Μαλή και εγκρίνει και την χρήση βίας και εδώ πρέπει να υπάρξει μια νέα σύνοδος για να υπάρξει απόφαση για τη μορφή που θα πάρει αυτή η αποστολή. Έχουμε και μια διπλωματική διαδικασία η οποία συνεχίζεται με διάφορες διαμεσολαβήσεις έχει επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή γιατί και η Βρετανία και η Αλγερία έχουν εμπλακεί πιο ενεργά μέσα σε αυτή τη διπλωματική διαδικασία και επιπλέον τίθενται τα θέματα της ασφάλειας με τις διάφορες εξελίξεις που έχουν λάβει η χώρα επιτοπίως με τις διάφορες ε, κινήσεις και κινήματα που έχουν κατακτήσει το Βόρειο Μαλί αλλά που είναι διχασμένες οι κινήσεις αυτές μεταξύ τους είμαστε και πάλι ενώπιον μιας κατάστασης η οποία είναι ιδιαίτερα ασταθής, αλλά χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση και έχει χρησιμοποιήσει τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Η Κατερίνα Άστον μας έχει υποστηρίξει πολλές φορές την ανάγκη μιας πλήρους και συνολικής ε, αντιμετώπισης και μετά από το κέρας της Αφρικής βλέπουμε ότι και στο Σαχέλ υπάρχει εύφορο έδαφος για να χρησιμοποιηθεί αυτή η συνολική αντιμετώπιση. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω καταρχής από τον κύριο Λόπεθ Μπλάνκο να μας κάνει μία επισκόψη των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Μετά ο κύριος Σαμπέρς για τα θέματα τα οποία είναι πιο λειτουργικού χαρακτήρα και μετά από τον κύριο Ντεκέρ για τις πτυχές ασφάλειας. Κύριε Λόπες. Ευχαριστώ κύριοι Ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ την ομάδα ΑΦΕΤ, την Επιτροπή ΑΦΕΤ, ε, για το ότι έβαλε το θέμα του Σαχέλ στην ημερήσια διάταξη και κυρίως το θέμα της κρίσης στο Μαλί. Θα μιλήσω τώρα στα αγγλικά, γιατί η παρουσίασή μου έχει ετοιμαστεί στα αγγλικά. Uh, Θέλω να σας ενημερώσω για την κατάσταση στην περιοχή, για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως ε, σε ό,τι αφορά τις ε, προκλήσεις ε, και την κρίση που προέκυψε μετά την κατάρρευση του κράτους στο Μαλί και να δούμε ποιες είναι οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ε, μακροπροθέσιμοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχά να προωθήσουμε τη σταθερότητα, να συνδέσουμε την ε, ασφάλεια, την ε, ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση, να υπάρχει συντονισμένη χρήση των εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζουν μια συνολική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουμε τις βαθιές αιτίες της έλλειψης ασφάλειας που οφείλονται στην περιφερειακή σύγκρουση και στα εθνικά προβλήματα ποια είναι η κατάσταση ασφάλειας και ποια είναι η πολιτική κατάσταση στο Μαλί. Η προετοιμασία της διεθνούς κοινότητας για να υποστηρίξει το Μαλί, ούτως ώστε να βοηθήσει το Μαλί να ανακτήσει την εδαφική του ακυρεότητα, έχει σημειώσει γοργή πρόοδο. Έγινε μια κοινή προσπάθεια επιχειρήσεων, ε, η Αφρικανική Ένωση, η Ευρωπαϊκή ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συμμετείχαν και στις 14 Νοεμβρίου η Αφρικανική Ένωση ενέκρινε τις προσπάθειες αυτές ε, και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα πάει στο τέλος του μήνα για να ετοιμάσει το δρόμο, ούτω ώστε να γίνουν συζητήσεις αρχές Δεκεμβρίου με σκοπό να υπάρξει ένα ψήφισμα υπό το κεφάλαιο 7, ε, ούτω ώστε η αποστολή, η οποία είναι διεθνής, αλλά υπό η αφρικανική αιγίδα για το Μαλί, ε, να λάβει την εντολή ούτως ώστε να αναπτυχθεί. Ε, κατά πάσα πιθανότητα αυτό το ψήφισμα θα εγκριθεί πριν το τέλος του 2012. Παρ' όλα αυτά, ε, σε πολιτικό επίπεδο δεν έχουμε κινηθεί επαρκώς. Ως πολιτική, οι πολιτικοί φορείς ε, εστιάζουν στην δημιουργία συνθήκων ε, με σκοπό να υπάρξει μια πολιτική μετάβαση παρά σε μια ε, συμφωνία για να αντιμετωπιστεί η θεσμική κρίση. Μέχρι στιγμής δεν έχει κινηθεί όσο θα έπρεπε η διεθνής κοινότητα. Δεν υπάρχει ένα αξιόπιστο πλαίσιο για διάλογο βορρά και νότου χωρίς τις τρομοκρατικές ομάδες για να επιληθεί η, κρίση στην οποία βεβαίως ε, συμμετέχουν και την προκαλούν και οι α, ε, τρομοκράτες. Η κυβέρνηση στην Παμάκο θα πρέπει να ενισχυθεί, να βοηθηθεί από τη διεθνή κοινότητα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Στο βορρά, ο χρόνος παίζει ε, υπέρ των Ισλαμικών ομάδων που είναι ένοπλες και ενισχύει το, την επιρροή που έχουν στο Βόρειο Μαλί και πάνω στον πληθυσμό, ε, οι οποίοι επιβάλλουν το νόμο της Αρία που παραβιάζει τα, τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, η Διεθνή τρομοκρατια τρομοκρατία ε, εμπνεύσεως Αλ-Κάιντα ε, ανθεί και βασιλεύει εκεί στο βόρειο ε, Μαλί και υπάρχει κίνδυνος για την πολιτική αστάθεια στις γειτονικές χώρες. Υπάρχει περίπτωση βέβαια να εξαπλωθεί η κατάσταση και το πρόβλημα και αλλού και στην Ευρώπη. Υπάρχει στρατολόγηση από τον ντόπιο πληθυσμό, υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ ένοπλων ομάδων το αποτέλεσμα των ε, διπλωματικών προσπαθειών της Αλγερίας και της Μπουρκίνα Φάσο καταγγέλλεται η τρομοκρατία στις 6 Νοεμβρίου έγινε αυτή η καταγγελία ε, γιατί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ε, την επιβολή του νόμου της Αρίας στο Βόρειο Μαλί. Επίσης ε, χρησιμοποιούν ε, αντάρτες του ΑΡΕΓ Ένας νέος γύρος συζητήσεων θα γίνει αρχές Δεκεμβρίου και αυτή την ε, φορά μπορούν, μπορεί να συμμετάσχουν και οι αρχές του Μπαμάκο με τη διαμισολάβηση της Μπουρκίνα Φάσο. Καλέ καλές είναι αυτές οι εξελίξεις, αλλά πρέπει να δούμε αν αυτή η νέα θέληση για διαπραγμάτευση με τον Μπαμάκο και με άλλες ομάδες είναι μια τακτική για να αποφευθεί η διεθνή στρατιωτική παρέμβαση ή απλώς ε, κερδίζουν χρόνο. Είναι σαφές ότι η διεθνής κοινότητα που προετοιμάζει τη στρατιωτική παρέμβαση αναγκάζει τους, ε, τις ένοπλες ομάδες να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ε, βέβαια αυτή τη στιγμή δίνουν διαβεβαιώσεις ότι θα κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και δέχονται μια ομοσπονδιακή λύση. Ε, οι ηγέτες παρόλα αυτά έκαναν μια στρατιωτική επιχείρηση ε, στα μέσα Νοεμβρίου. ούτω ώστε να έχουν περισσότερα χαρτιά στο χέρι τους εν ώψη των ε, επερχόμενων διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ αυτές οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει και απώλειες αμάχων. Το MNLA στο μεταξύ συμπίζει συμμαχίες με διάφορες άλλες ομάδες. Ποιοι είναι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπό έχει καταρχήν να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της ε, διαδικασίας μετάβασης με σαφείς προθεσμίες, ούτως ώστε να υπάρξει μια εκλεγμένη κυβέρνηση που να ασκήσει πραγματικό έλεγχο και να βοηθήσει στην δημιουργία ενόπλων δυνάμεων. Ε, υπάρχει πρόγραμμα ε, συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την εφαρμογή του οδικού χάρτη που έχει τους στόχους που σας προανέφερα. Επίσης να υπάρξει ένα πραγματικό πλαίσιο για διάλογο βορρά και νότου, ε, ούτως ώστε οι παραδοσιακοί ηγέτες ε, να συμμετάσχουν στις ειρηνευτικές συνομιλίες, ε, χωρίς τη συμμετοχή των ε, ηγετών των τρομοκρατικών ομάδων. και να αναπτύξουν δραστηριότητες διαμεσολάβησης βάσει του επίπεδου track 2 και track 3. Τέταρτον, θα πρέπει να γίνει πιο ε, ισχυρή η απειλή βίας για να μπορέσουν να προωθηθούν οι διαπραγματεύσει και τέλος για να χρησιμοποιηθεί βία κατά των τρομοκρατών και των εγκληματικών ομάδων εάν αυτό είναι απαραίτητο. Αυτή είναι η γραμμή που έχει ακολουθήσει η ΕΟΚΑΠ, η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ήγερα και αυτή θα είναι η γραμμή που θα ακολουθήσει η αποστολή αυτή της ΚΕΠΑ στην περιοχή. Τέταρτον, θα πρέπει να επαναφέρουμε την αξιοπιστία του, των κρατικών δομών και να επαναφέρουμε το κοινωνικό συμβόλαιο. ώστε να προκύψει και το λεγόμενο μέρισμα ειρηνη εάν υπάρξει συμφιλίωση. τέλο. θα πρέπει να υποστηρίξουμε την σταθεροποίηση, την συμφιλίωση και την οικοδόμηση τη ειρήνη στον Βορρά με το ενδεικτικό πρόγραμμα το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι χρειάζονται κατεπίγοντα μέτρα και δεσμεύσει σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Θα σα κάνω τώρα μια σύνοψη των δραστηριοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταλήξω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία της, της στρατηγικής του Σαχέλ. Έχει υπάρξει έντονη διπλωματική δραστηριότητα η οποία έχει αποδώσει καρπούς και εκεί περιλαμβάνω και τις ενέργειες του κυρίου Ζιλντε Κερκόβ, ο οποίος είναι ο συντονιστής για τα αντιτρομοκρατικά θέματα. Αυτή η δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναγνωριστεί σε όλα τα διεθνή φόρουμ και η στενή συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση και τον ΟΗΕ είναι πολύ θετική. Με τον τρόπο αυτή η στατιωτική επιχείρηση της ΚΕΠΑ έχει σαν στόχο την κατάρτιση και την αναδιοργάνωση του Μαλιανού στρατού και δεν έχει προσκλούσει σε καμία επιφύλαξη από τις αρχές του Μπαμάκο, που είναι οι νόμιμες αρχές της ε, χώρας αυτής του Μαλή. Θα είναι ένα κομβικό στοιχείο της ε, δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Έχουμε σαν στόχο από τη στιγμή που θα υπάρξει το απαραίτητος, ο απαραίτητο οδικό χάρτη να επαναλάβουμε τι δράσει ανάπτυξη για να υποστηρίξουμε και τι κινήσει προ μια πολιτική μετάβαση οι προσπάθειες διαμεσολάβησης υποστηρίζουν τους τοπικούς και διεθνείς διαμεσολαβητές ώστε να προκύψει μια πλήρης λύση. Τέλος, χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για να ενισχυθεί και η σταθερότητα των ομόρων χωρών, ιδίω μέσω της αποστολής ΕΟΚΑΠ, για την οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Στη Μαυριτανία, οι χώρες αυτές οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως η Μαυριτανία, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ανθρωπιστικές και πτυχές ασφάλειας για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε και παραμένω στη διάθεσή σας για όλα τα θέματα που θελήσετε εγείρη. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που θέλουν να υποβάλουν συνάδελφοι. Που το, το λόγο έχει πρώτα ο κύριος ε, Αμπέρ. Πρόκειται για αυτή τη νέα αποστολή στον ε, Νίγερα και για την προετοιμασία συνακόλουθα της αποστολής στο Μαλί. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου. Όπως είπε ο κύριος Λόπες Μπλάνκο, η αποστολή στον ε, Νίγηρα ε, προχωρεί και συνεχίζει να εξελίσσεται. Πρόκειται για απόφαση Συμβουλίου του 16 Ιουλίου. Ε, αφορά περίοδο διετή με προσωπικό 50 πρόσωπα των επικεφαλής είναι ο Φρανσίσκο Σπινόσα της Ισπανικής Guardia Civil που είναι ο επικέφαλή της αποστολής και πρόκειται για αποστολή εκπαίδευσης και παροχή συμβουλών αποσπασμένοι ε, υπάλληλοι από, από αστυνομία, στρατό και ο καθένας λοιπόν στον τομέα του θα βοηθήσει όσον αφορά την ασφάλεια του Νίγηρα. Ο επικεφαλής της αποστολής επομένω έχει μαζί του μια ομάδα 25 οι οποίες στο DMA αναπτύχθηκαν στις 8 8 και στην ΙΑΜΗ ακόμα βρίσκονται αυτοί οι 25 μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου η αποστολή θα φτάσει στους 45 με 50. Στις 10 Δεκεμβρίου ο επικεφαλής της αποστολής πρόκειται να υποβάλει στο ΣΥΦΚΟΜ τα σχέδιά του, το, το πρόγραμμά του και δεν νομίζω να υπάρχουν τίποτα μείζονες αλλαγές σε σχέση με, την, ε, με τις αρχικές κατευθυντήριες. Οι στόχοι της αποστολής είναι παροχή συμβουλών, αρρωγή όσον αφορά την ασφάλεια της στρατηγικής της χώρας για ανάπτυξη και θα βοηθήσει όσον αφορά κάποιον συντονισμό περιφερειακό και ευρύτερο και να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία. Να ενισχυθεί το κράτο δικαίου μέσω αναβάθμισης ε, των ε, ανακριτικών και λοιπόν ποινικών διαδικασιών to support the development of the Nigerian security forces and to contribute Βοήθεια στις, ε, στις αρχές, προγραμματισμός, υλοποίηση προγραμμάτων, σχεδίων όσον αφορά πάντα την ασφάλεια. Όπως προανέφερα, η αποστολή αυτή ξεκίνησε, πάντων αποφασίστηκε να γίνει στις 16 Ιουλίου. Ο δε επικεφαλής είπαμε ότι μετέβη στις 8-8 με την ε, ομάδα του, με το επιτελείο του. Αλλά η αποστολή ακόμη δεν έχει υποβάλει το επιχειρησιακό σχέδιο. Αυτό το οποίο καθορίζει κάθε κίνηση. Όμως, ήδη έχουν γίνει επαφές με τους τοπικούς παράγοντες στον τομέα της ασφάλειας του Νίγηρος. να έχουν γίνει σωστέ διασυνδέσει, αλλά ακόμα δεν έχει αρχίσει η υπηρεσιακή δραστηριότητα πλήρω. Και γιατί αυτό, γιατί υπάρχουν συνήθεις δυσκολίες. Ότι το σύμπησε εσύ. Θέλουμε να υπάρχει αυτή τεχνική μελέτη και να πάμε να δούμε, να διερευνήσουμε υπό ποιου ορους και προποθεσεις ε, εξελίσσεται αυτή η αποστολή. Αλλά τα σχετικά κονδύλια θα εκταμιευτούν μόλις επισημοποιηθεί ή ο διορισμός του επικεφαλής επομένως διαδοχικά εκεί έγιναν τρεις αποστολέ. Και τρεις επομένως θα έπρεπε να έχουν αυτάρκεια και αυτοδυναμία. Βεβαίω και η αξιολόγηση της ασφάλειάς τους πρέπει να γίνεται, κάτι το οποίο είναι βασική μας μέρημνα και στον Νίγηρα. Θα έπρεπε ο, ο καθένας να βρει τα, τα τηλέφωνα και λοιπόν υλικό επικοινωνία και μέσα επικοινωνία. Αυτό δεν είναι τόσο θέμα υλοποίησης εντολής. Είναι θέμα των συνθήκων, προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν για να πετύχει αποστολή. Επίση. έχουμε προβλήματα όσον αφορά την επάνδρωση του, της αποστολής, γιατί όλοι όσοι συμμετέχουν σε αποστολή δώσανε συνέντευξη, αλλά δεν είχαμε ε, τη δυνατότητα να, να κάνουμε σε, σε, σε, ένα συγκεκριμένο, σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα τις 100 περίπου συνέντευξη που χρειάστηκαν. Οπότε γι' αυτό το λόγο κάπου υπήρξε εμπλοκή και στον Ήγηρα, αλλά και στις άλλες αποστολές. Καφές και άλλο και άλλο στην Αφρική. Και στο Νότιο Σουδάν, για να μην πούμε τι γίνεται και στις άλλες αποστολές, είχαμε αντικαταστάσεις προσωπικού και σε σχέση με τις συνεντεύξεις, γιατί επίσης στις 10-12 του πρόκειται να γίνει παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου. Οπότε και τότε θα ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις. Οπότε νομίζω την επόμενη φορά θα συζητήσουμε πιο ουσιαστικά πράγματα. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντεκέρκοφ. Όπως ε, ήθιστε θα προβεί σε μια αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας σε σχέση με τις διάφορες ε, με ομάδες και τα διάφορα κινήματα τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή αυτή και θα μπορέσουμε στη συνέχεια να σταθούμε περισσότερο στις περιφερειακές απειλές γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί δεν είναι απομονωμένα και έχουν επιπτώσεις και στην περιραίουσα περιοχή. Σας ευχαριστώ για την ε, προσοχή που έχετε δώσει για το θέμα αυτό. Και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η περιοχή και συμφωνούμε για την ε, ασφάλεια και της ίδιας της Ευρώπης. Όπως είπατε, δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο για το Μαλί. Έχει χάσει την εξουσία πάνω στα δύο τρίτα του, της επικράτειάς της στο κυβέρνηση του Μαλί, που είναι τώρα ασφαλές καταφύγιο για ε, πολεμιστές του Ισλάμ και που αρχίζουν να αποσταθεροποιούν και τις όμορες περιοχές. Δεν είναι μόνο ο αντίκτυπο για τον Ήγερα και τη Μαυριτανία που προκύπτει από αυτές τις ενέργειες, αλλά και ο κίνδυνος να αποσταθροποιηθεί και η Σενεγάλη, το Μπουρκίνα Φάσο, ακόμα και το Τσάντ. Βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει αυτή η διείσδυση και η επιρροή αυτών των τρομοκρατικών ομάδων στους καταβλισμούς ε, προσφύγων, όπου υπάρχουν ε, πολλοί άνθρωποι στο Μαλί. Και είδαμε επίσης και στο Τιντούφ στην Αλγερία, στον καταβλισμό των ε, Σαχαραουί, να υπάρχει σημαντικός αντίκτυπος γιατί υπήρξε απαγωγή πολλών και υπήρξαν και κάποιοι Σαχαρούι οι οποίοι πήγαν να συνταχθούν με τους τρομοκράτες στο Μαλί. Υπάρχει λοιπόν αντίκτυπος και στο Βορρά και στο Νότο. Είδαμε στη Βενγκάζη, στη Λιβύη ότι οι συνεργάτες των ε, Μαλιανών δεν είναι αδρανείς, υπάρχει παρουσία λοιπόν αυτών των οργανώσεων και στη Βόρεια Λιβύη, αλλά υπάρχει και διείσδυση προς την κατεύθυνση της Τινησίας, και στο Μαρόκο υπάρχει μεγάλη ανησυχία γιατί υπάρχουν πολλοί νέοι Μαροκινοί οι οποίοι φεύγουν από το Μαρόκο για να καταταγούν σε αυτές τις ομάδες. Ο κίνδυνος είναι ότι θα επανέλθουν και θα ε, κάνουν τρομοκρατικές ε, δράσεις. Η ΑΚΙΜ λοιπόν, η ΑΚΜΗ είναι αυτοί <clears throat> οι οποίοι ε, εκπαιδεύουν πολλούς από το Μπόκο Γαράμ στην Ιγυρία και υπάρχει ο κίνδυνος εν καιρό ότι θα υπάρξει μια συνεργασία της Al-Shabaab, του Ακμή και του Μπόκο Χαράμ. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ανησυχητικό σενάριο για την ανάπτυξη και την μελλοντική εξέλιξη στην Αφρική. Όλα αυτά γίνονται με βασικό καμβά επίσης μια έκρηξη της χρήσης και εμπορίας ναρκωτικών. Ακόμα και αν υπάρχουν πολλές συζητήσεις μεταξύ των υπηρεσιών ασφάλειας για το αν η ΑΚΜΗ ε, εμπλέκεται σε αυτήν την διαδικασία, <clears throat> είναι φανερό ότι υπάρχουν τμήματα αυτής της οργάνωσης που ενδεχομένως να ασχολούνται με την κυκλοφορία ναρκωτικών. Υπάρχει πάντως μια έκρηξη της κυκλοφορίας ναρκωτικών στη Δυτική Αφρική και ξέρουμε πώς τα ναρκωτικά καταστρέφουν την ευκυβερνησία. Υπάρχουν πολλά κράτη λοιπόν τα οποία είναι εύθραυστα και μπορούν να αντιμετωπίσουν ανάλογες κατάστασης. Αυτά λοιπόν για την περιοχή. Για μας τώρα ως Ευρωπαίους έχουμε αρχίσει να βλέπουμε, αλλά δεν έχουμε ακόμα σημαντικά στοιχεία. Αρχίζουμε να βλέπουμε ένα αριθμό νέων που έχουν πολλές φορές διπλή υπηκότητα, διπλά διαβατήρια, να πηγαίνουν στην περιοχή αυτή. Υπήρξαν κάποιες συλλήψεις στη Γαλλία και στο Βέλιο. Υπάρχουν οι Γερμανοί, Αυστριακοί, ε, υπήκοοι που βρίσκονται στα στρατόπεδα της Λιβύης και οι οποίοι είναι έτοιμοι να ε, συνενωθούν με τις διάφορες εγκληματικές οργανώσεις στο Μαλί. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα αυτό. Όπω είπε και ο κύριο Λόπε, μπορούμε να εκφράσουμε την καροποίησή μα για το γεγονό ότι η διεθνή απάντηση και ιδίω η απάντηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στεναρή και ισχυρή. Και αναπτύσσουμε το πλήρε φάσμα των εργαλείων που έχει στη διάθεσή τη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από 3-4 χρόνια ακολουθούσαμε την κλασική οδό ενίσχυσης ικανοτήτων με εργαλεία σταθερότητας, επιδοτήσεις από την πλευρά του, του Ταμείου Ανάπτυξης. Σήμερα αρχίζουμε να εμπλεκόμαστε περισσότερο με αποστολές πολιτικού και στρατιωτικού χαρακτήρα, την ΕΟΚΑΠ στο Νίγηρα και την αντίστοιχη αποστολή στο Μαλί. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, γιατί όσο καθυστερούμε τόσο αυτές οι τρομοκρατικές ομάδες ενισχύουν τις ρίζες που έχουν στην περιοχή αυτή. Σήμερα δεν μπορούν στο Βόρειο Μαλή να εισέλθουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και είναι σαφές ότι η τροφοδοσία σε τρόφιμα και σε, φάρμα, σε φάρμακα, η διαχείριση καθημερινής ζωής, όλα αυτά βρισκόνται στα χέρια των τρομοκρατών. Δεν είναι, υπάρχει αμφιβολία ότι όταν ελέγχετε την καθημερινή ζωή, μπορείτε να στρατολογείτε και νέους από τις οικογένειες της περιοχής. Είναι λοιπόν σημαντικό. Να ετοιμαστούμε και οι αποστολές αυτές να, να αναπτυχθούν το συντομότερο δυνατό. Όσο πιο γρήγορα παρέμβουμε, καλύτερα θα είναι. Όχι μόνο τεχνικός πώς, αλλά και γιατί η πίεση, η στρατιωτική πίεση βοηθάει παραδόξως τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για τις οποίες μίλησε ο Μανουέλ. Χαίρομαι λοιπόν που επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί χρειάστηκε χρόνο για να κουνηθεί, ε, τελικά ε, συμφώνησε, συμφώνησαν τα 27 κράτη-μέλη, ούτως ώστε ε, να αναπτύξουν όλα τα μέσα για να αναπτυχθεί αυτή η επιχείρηση στο Μαλί. Εδώ και δύο-τρία χρόνια εγώ πίεζα. Επομένως, το μήνυμά μου σήμερα είναι το εξής. Είμαι θειασότης πραγματικά αυτής της ε, αποστολής, ε, αυτής της επιχείρησης της ΚΠΑ. Και λέω ότι αυτή η αποστολή δεν πρέπει να είναι, αυτή η επιχείρηση δεν είναι η μόνη απάντηση. Ο Μανουέλ Λοπέζ ε, μιλά για μια συνολική σφαιρική στρατηγική, δηλαδή να καλύψουμε όλες τις πτυχές, την πρόληψη, τη διακυβέρνηση, την ανάπτυξη, ε, να αντιμετωπίσουμε επίσης τη ριζοσπαστικοποίηση. Μην πιστεύετε ότι επειδή έχω μια επιχείρηση ε, 300 ας πούμε ε, στρατιωτικών τέλειωσε το θέμα. Πολλά ακόμα πράγματα πρέπει να γίνουν, ε, ιδίω ε, στην αντιτρομοκρατία, εκεί όπου είμαι υπεύθυνο εγώ. Ε, και θα σας δώσω κάποιες ιδέες για το τι πρέπει να κάνουμε πάρα αυτά σήμερα, τώρα, παράλληλα με τις στρατιωτικές προσπάθειες θα σας πω για, τι πρέπει να κάνουμε για την πρόληψη, για την ασφάλεια, για τον ανεφοδιασμό, ούτω ώστε να παρεμποδίσουμε τον ανεφοδιασμό των τρομοκρατικών ομάδων μέσω των, του γαθρεμπορίου. Ε, και τι μπορούμε να κάνουμε για τις όμορες χώρες, ε, Νίγηρο, Μαλή και Μαυριτανία. Σε ό,τι αφορά την πρόληψη, ε, μπορούμε να κάνουμε πολλά. Είναι κρίσιμος τομέας, αλλά δύσκολος παράλληλα. Έχουμε υπάρχει ένας αντίλογος. Μπορούμε δηλαδή να αναπτύξουμε έντονες δράσεις ε, που δημιουργούν άλλη νοοτροπία ε, στην, ε, στην περιοχή. Όταν βλέπουμε, ας πούμε, την συμπεριφορά αυτών των τρομοκρατικών ομάδων, του ΑΚΙΜ και τα λοιπά, έχουν επιβάλει την, το Σαρία, αλλά με φοβερά βίο τρόπο. Με λιθοβολισμό, με απίστευτα βασανιστήρια, με δολοφονίες, βιασμούς, ε, στρατολόγηση παιδιών στρατιωτών και λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Έχουμε Καλό είναι να έχουμε λοιπόν, έχουμε μάλλον αυτές τις ομάδες που κάνουν ακριβώς το αντίθετο από το Ισλάμ που θέλουν να προωθήσουν. Εμείς θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Στο Αλγέρι υπάρχει και ένα κέντρο που δημιούργησε η Αλγερία και οι τρεις όμορες χώρες ούτω ώστε να συλλέξουν πληροφορίες και είναι ένας πυρήνας παράλληλα, ο οποίος ε, δουλεύει πάνω σε θέματα πρόληψης. Και ένα από τα προγράμματα που κάνει προσπαθήσει να μοιράσει ε, ραδιόφωνα τα οποία λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, ούτω ώστε να προωθήσουν τι αντίθετε ιδέε και να δείξουν την πραγματικότητα, να εκμεταλλευτούν τη βία και το πρόβλημα που υπάρχει, α πούμε, για να καταλάβει ο κόσμο και να το κατανοήσει. Το πρώτο που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να υποστηρίξει τέτοια προγράμματα. Δεύτερον, ε, δεν θα κάνω σύγκριση τώρα με το Αφγανιστάν, γιατί είναι απλοϊκό να μιλάμε για ταλιμπανισμό και αυγανοποίηση κτλ. Αλλά αυτό που μάθαμε από την παρέμβασή μας στο Αφγανιστάν είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε και σε στρατιωτικό και σε πολιτικό επίπεδο παράλληλα. Και το, αυτό που λέμε ε, καθαρίζουμε, κρατάμε και χτίζουμε τι σήμαινε ουσιαστικό το Γκάο ή την Μπουκτού. Έχει νόημα να τις ε, καταλάβουμε αυτές τις πόλεις, αλλά, αλλά παράλληλα και όχι έξι μήνες μετά. Αν δεν δώσουμε μια πολιτική απάντηση στις προσδοκίες του πληθυσμού, όχι μόνο αυτοί οι πληθυσμοί δεν θα πιστούν για την παρέμβασή μας, αλλά θα παραμείνει ο κίνδυνος οι νέοι, οι κάτοικοι να προσφύγουν σε αυτές τις τρομοκρατικές ομάδες. Όταν ξέρουμε την φοβερή αργοπορία της ανάπτυξης τέτοιων αναπτυξιακών προγραμμάτων, ε, ήδη από σήμερα πρέπει να ξεκινήσουμε να ετοιμάζουμε μια πολιτική απάντηση, ούτω ώστε παράλληλα με τη στρατιωτική ενέργεια, όταν καταλάβουμε αυτές τις τρεις πόλεις και τη γύρω περιοχή, να έχουμε έτοιμη μια μη στρατιωτική απάντηση. Ε, στο Βόρειο Μαλί προσπαθούμε να υποστηρίξουμε ένα σχέδιο που είχε ε, ετοιμάσει ο πρόεδρος, δηλαδή ε, γύρω από τι στρατιωτικέ βάσει να υπάρχουν ε, κοινωνικέ υπηρεσίε, να αρχίσει να αναπτύσσεται ένα κράτο. Αλλά δεν υπήρχε αρκετή πολιτική συνένεση. Δεν υπήρχε αρκετή θέληση ούτε μέσα ούτε εξήγηση στον πληθυσμό. Θα πρέπει όμω κάτι τέτοιο να προωθήσουμε, αν όχι αυτό. Τρίτον, επίση θα πρέπει να εξηγήσουμε κάτι πολύ συχνά ο Μανουέλ. Όταν ξέρουμε την ε, κοινωνία στο Μαλί, δεν είναι σίγουρο ότι όλοι στον Παμάκο είναι πεπισμένοι ότι οι εχθροί είναι οι τρομοκράτες. Υπάρχει μια τεράστια δουλειά συμφιλίως πρέπει να κάνουμε ανάμεσα στους Τουαρέ και στον πληθυσμό του Μαλή. Θα πρέπει λοιπόν να εξηγήσουμε στον πληθυσμό του Βορρά γιατί κάνουμε μια στρατιωτική παρέμβαση, αλλιώ, δεν περνάει το μήνυμα. Ε, το ίδιο πρόβλημα που θα έχουμε και στο Αφγανιστάν. Τέταρτον, δικαιοσύνη. Θα υπάρξει ε, μία μη διεθνής ε, στρατιωτική ε, παρέμβαση ε, για να σταματήσουμε τους τρομοκράτες. Κάποιους θα τους σκοτώσουμε. Κάποιοι θα σκοτωθούν. Ε, θα πρέπει μετά όμως να περάσουμε και σε επίπεδο δικαιοσύνης. Δεν είναι σίγουρο ότι οι αρχές του Μαλή σήμερα είναι σε ε, θέση να διαχειριστούν ένα πακέτο κρατουμένων για, που είναι κρατούμενοι για λόγους τρομοκρατίας. Επομένως, μόλις θα επιτρέψει η πολιτική κατάσταση θα πρέπει να ενισχύσουμε την ικανότητα της κυβέρνησης του Μαλή να δώσει μια δικαστική απάντηση. Σίγουρα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ίσως ας πούμε, διερευνήσει κάποια εγκλήματα, αλλά θα πρέπει η πολιτική δικαιοσύνη να το κάνει, η μη στρατιωτική. Ο συνάδελφος του CPCC θα σας μιλήσει για αυτά, αλλά η κατάρτιση, η εκπαίδευση του στρατού του Μαλή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το σεβασμό των ανθρωπιστικών δικαιωμάτων ε, για να μην υπάρχουν διολυστήσεις. Επίσης, η πρόληψη στο νότιο Μαλή, άλλο στοιχείο. Αν κοιτάξετε την εξέλιξη της ε, κοινωνίας του Μαλή, ε, εξελίσσεται όπως η κοινωνία στη Μαυριτανία πριν από 10 χρόνια. Δηλαδή μια Ισλαμοποίηση τρομακτικά γρήγορη στην κοινωνία αυτή, με μια όλο και μεγαλύτερη ε, επιρροή. Αν κοιτάξετε, ας πούμε, το Ανώτατο Συμβούλιο, το Μουσουλμανικό στον Παμάκο, έχει μια φοβερή επιρροή που δεν είναι το παραδοσιακό Ισλάμ. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια προσπάθεια και στο επίπεδο της πρόληψης. Ε, το επόμενο, ε, τα στρατόπεδα προσφύγων. Θα ήθελα η Κομισιόν και υπάρχουν κάποια προγράμματα που έχουν τρομολογηθεί να δώσουν προσοχή ε, στα στρατόπεδα προσφύγων στη Μαυριτανία, στον Ήγυρα, ε, στους Σαχαράουι. Υπάρχουν εκεί νέοι, άεργοι, ε, έφηβοι που δεν έχουν καμία εκπαίδευση, που είναι ένα απίστευτο φυτόριο για να στρατολογηθούν, ας πούμε, τρομοκράτες για αυτές τις ομάδες. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε πάρα αυτά. Τελευταίο στοιχείο είναι η διαμεσολάβηση. Το Μανουέλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να υποστηρίξει την διαμεσολάβηση της Μπουρκίνα, Φάσο. Υπάρχουν και διάφορες ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις που δραστηριοποιούνται. Αν να γίνει κάτι τώρα πρέπει να το κάνουμε. Ε, μαζί με την αξιόπιστη στρατιωτική απειλή θα πρέπει να προσπαθήσουμε α, όλους αυτούς που πήγαν σε αυτές τις τρομοκρατικές ομάδες για οικονομικούς λόγους, έτσι από οπορτονισμό ας πούμε, και που δεν ε, συμμερίζονται την ιδεολογία, να τους αποσπάσουμε από εκεί. Αυτά για την πρόληψη. Στον τομέα της ασφάλειας. Εγώ κάνω έκκληση να στείλουμε ήδη από σήμερα, να ασχοληθούμε μάλλον με τον Ήγηρα, ε, να ξεκινήσει αυτή η αποστολή ΕΟΚΑΠ στον Ήγηρα. Δεν έχουμε αρκετό προσωπικό και να αναπτυχθεί και στο Μαλί και στη Μαυριτανία. Γιατί να περιμένουμε ακόμα ένα χρόνο, δεν το καταλαβαίνουμε, ούτω ώστε ε, να αναπτύξουμε αυτήν την αποστολή ΕΟΚΑΠ που θέλει να δώσει κατάρτιση στους αστυνομικούς, ε, στους δικαστικούς. Είναι σημαντικό και για το Μαλί και για τη Μαυριτανία και για τον Νίγηρα. Κάτι άλλο πιο εσωτερικό τώρα. Ε, δουλέψαμε, ε, όχι ε, με σταθερότητα. Ε, δουλέψαμε βαθμιδών. Ε, ξεκινήσαμε από προγράμματα επιδοτήσεων. ένα πρόγραμμα 6,5 εκατομμυρίων στην αρχή, με σκοπό την, το νόμο και την τάξη. Και μετά προσθέσαμε την ΕΟΚΑΠ με το ίδιο θέμα. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν να προχωρήσουμε, να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας και υπάρχουν διάφορα κρατημέλη, ιδίω η Γαλλία και κάποια άλλα όμω, που προσπαθούν να αναπτύξουν τη δικαιοσύνη στι χώρε του Σαχέλ. Υπάρχει μια κουλτούρα όμω ατιμορρησία η οποία είναι τεράστια, τόσο σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία όσο και την ναρκωτικά. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό. Θα πρέπει να μπορούμε να στέλνουμε το μήνυμα ότι το έγκλημα οδηγεί σε τιμωρία, στη φυλακή. Άμα δεν τα καταφέρνουμε. Γιατί το ε, λαθρεμπόριο διαφύρει. Γιατί όχι. Να δημιουργήσουμε ένα περιφερειακό μηχανισμό διώξεων των μεγάλων λαθρεμπόρων Επιπλέον, τα σύνορα. Εσάς έχω δουλέψει πάνω στα σύνορα όταν ασχολήθηκα με την Αλγερία. Θα πρέπει να γίνει μια, μια μεταρρύθμιση ε, στα σύνορα καταρχάς στα σύνορα της, της Λιβύης, στα πλαίσια των, ε, της κατανομής ε, των αρμοδιοτήτων στον, ΟΗΟ, στον ΟΗΕ, ε, θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει γενικά μετά τα σύνορα των χωρών Σαχέλ. Μπορεί κάποια στιγμή να παρεύουμε στην ε, Λιβύη με μια αποστολή ΚΠΑ, θα πρέπει να δούμε και τα σύνορα γενικά στη Σαχέλ. Τώρα για τη Μαυριτανία έχουμε 20 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για να βοηθήσουμε την άμυνα αλλά και τη δικαιοσύνη και την αστυνομία. Θα πρέπει να επιταχύνουμε αυτά τα προγράμματα και σε εσωτερικό επίπεδο έρχομαι σε επαφή με τους συναδέλφους που ασχολούνται με τη δικαιοσύνη και τα εσωτερικά και με τις υπηρεσίες Europol, Eurojust κτλ. ώστε να δουλέψουμε πιο ενεργά για τον έλεγχο και την πρόληψη των ε, τζιχαντιστών Τη Ευρώπης που θέλουν να πάνε να μεταβούν εκεί στο Σαχέλ. Επίσης, ε, το θέμα του ανεφοδιασμού. Αν κοιτάξετε την ΑΚΙΜ, έχουν λεφτά από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Ε, καλά είναι τα λεφτά, αλλά πρέπει να τα μπορούν να χρησιμοποιούν. Πρέπει να ανεφοδιαστούν ε, σε ανταλλακτικά, σε ε, βενζίνη, τρόφιμα κτλ. Και ξέρετε πολύ καλά ότι η οικονομία του Βορείου Μαλή είναι στραμμένη πιο πολύ προς την Αλγερία παρά προς την πρωτεύουσα του Μαλή του Μπαμάκο. Ε, είναι πολύ συνδεδεμένη με την Αλγερία λοιπόν. Ε, είναι λοιπόν πολύ πιο σημαντικό να συνεργαζόμαστε με τους Αλγερινούς. Εντάξει, είναι δύσκολο να ελέγξουμε ε, τα σύνορα στην ε, ε, έρημο. Αλλά οι Αλγερινοί ξέρουν πολύ καλά να ελέγχουν τα σύνορά τους. Παρά να προσπαθούμε να κλείσουμε τα σύνορα του Μαλή. Το επόμενο, ναρκωτικά. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Με κατάπληξη άκουσα ότι η ειδική υπηρεσία του ΟΗΕ για τα θέματα ναρκωτικών θα κλείσει το γραφείο της στη Γουινέα Μπισάου που είναι η μεγαλύτερη χώρα λαθρεμπορού ναρκωτικών στον κόσμο. Δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να έχει γραφείο αυτή η υπηρεσία, είναι εκεί πέρα. Και γιατί, γιατί δεν έχουν λεφτά τα κράτη-μέλη. Μα δεν έχει νόημα, είναι παράλογο. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα από αυτά. Ε, στα θέματα δικαιοσύνη εσωτερικών υποθέσεων θα πρέπει να προωθήσουμε διάφορα ε, προγράμματα στον Τακάρ, στην Άκρα κτλ. Στη Τουλόν. Επίση, συνεργαζόμαστε με την Ιντερπολ. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Υπάρχουν δύο ιδέε ε, που μπορεί ίσω να εφαρμόσουμε, αν και είναι δύσκολε. Ε, Πρώτον, ένα ε, περιφερειακό μηχανισμό διώξεων των ε, μεγάλων λαθρεμπόρων, γιατί υπάρχει πολλή πίεση στου δικού μα δικαστέ. Ε, υπάρχουν πολλά χρήματα που κυκλοφορούν. Και επίση, γιατί να μην διαρευνήσουμε στον ΟΗΕ ε, τη δυνατότητα ύπαρξη ενό μηχανισμού κυρώσεων ε, εναντίον των λαθρεμπόρων ναρκωτικών. Το κάναμε για του τρομοκράτε. Ούτω ώστε στην Δυτική Αφρική, που για τη Δυτική Αφρική μάλλον είναι απειλή για την ασφάλεια και την ειρήνη. Και τελευταίο πράγμα, ο δεύτερος κύκλος όπως είπα, ε, ανησυχούμε τι επίπτωση θα έχουν όλα αυτά στους γείτονες Σενεγάλη, Μπουρκίνα Φάσο. Χρήσιμο λοιπόν θα ήταν να διερευνήσουμε και εκεί τι μπορούμε να κάνουμε παραπέρα. Ε, ο πρόεδρος της Σενεγάλης ήρθε εδώ στις ε, Βρυξέλλες και μας ρώτησε τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο ασφάλειας. Θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε τις ανάγκες τους και να κινητοποιήσουμε περισσότερα μέσα από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, ούτως ώστε να μην ξανάρθουμε εδώ αύριο και συζητάμε τι δεν πήγε καλά στη Σενεγάλη. Πρόληψη καλύτερη από τη θεραπεία. Αυτή είναι κάποιοι τομή που πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερο. Παράλληλα με αυτή την παράλληλη ανάπτυξη της στρατιωτικής αποστολής στο Μαλί που πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την τόσο άρτια σύγχυση η οποία περιείχε όλες αυτές τις ε, ιδέες μας τα είπατε τόσο συγκεκριμένα και τώρα που σας ακούω να σας πω τι, τι, τι μου ήρθε στο μυαλό. Όχι δεν φταίτε εσείς, αλλά θεωρώ ότι χάθηκε πολλής χρόνος γιατί τόσα χρόνια χτύπαγε το καμπανάκι ο κόδων κινδύνου για αυτή την περιοχή, για το Σαχέλ. Και βεβαίω πρόκειται για όλε αυτέ τι θετικέ προσπάθειε και νομίζω ότι είναι σαφέ ότι συμφωνούμε ότι τέτοιε ε, αποστολέ πρέπει να γίνονται εδώ στο Κοινοβούλιο. Αλλά παρόλα αυτά, η εντύπωσή μου είναι ότι η προσπάθεια τώρα έφτασε να γίνει αργά. Ε, λέμε τώρα για, για, εκπαίδευση, κατάρτιση και όλα αυτά, ενώ το, το, το πρόβλημα έχει παρεξενθεί και από ό,τι φαίνεται οι χώρες της περιοχής αυτής τώρα μετά την διπλωματική πίεση που ασκήθηκε σε σχέση με την στρατιωτική επανέβαση, περισσότεροι λοιπόν εκεί πέρα και οι διαμεσολαβητέ, ακούσαμε τι είπε και ο πρώτη, επιμένουν, επιμένουν πολύ τώρα όσον αφορά την πολιτική και διπλωματική διάσταση του προβλήματος. Άρα μάλλον βασιλεύει σύγχυση. Και από την άλλη μεριά έχουμε αυτή την μεγάλη καθυστέρηση, μια στρατηγική η οποία επί 1,5 χρόνο είχε μπλοκαριστεί και θα πρέπει να έχουν γίνει όλα αυτά πιο νωρί. Βεβαίω ε, δεν είμαι αφελή. Ξέρω ότι όλα εξαρτώνται από το ρυθμό απόφαση του Συμβουλίου. Πρόκειται για το πόσο ευαίσθητα είναι τα, τα, τα Δεν έχουν όλοι την ίδια αντίληψη και ευαισθησία για το πρόβλημα. Οπότε βεβαίω Εντάξει, κρούσατε τον κόδωνα του κινδύνου, σωστό, αλλά τέλο πάντων. Ε, να δούμε τώρα τι ερωταπαντήσει του υποφαινομένου αλλά και των συναδέλφων και σε σχέση με τι αρμοδιότητέ σα, σε σχέση με τη δομή που έχει ο φορέα σα, το, σώμα αυτό το οποίο γίνεται, για πετε μα, τι λέτε εσεί για, για, αυτή την καθυστέρηση. Να, συγκεκριμένο, τι γίνεται σε σχέση με την ε, αποστολή στον Νίγηρα. Έχουμε την απόφαση του Ιουλίου για τον Ήγηρα, οπότε και εδώ πέρα πάλι κολλάμε στα ίδια και στα ίδια σε σχέση με αυτές τις αποστολές γιατί ακριβώς ε, είπαμε ότι ε, ε, δεν έχουμε 2.000 άτομα να στείλουμε, στείλαμε στο Κόσοβο. Έχουμε μόλις 50 άτομα, όμως παρόλα αυτά έχουμε προβλήματα υλικά, χρηματοδότησης, δεν έχουν καν, καν, καν να τους δώσουν. Ο, ο καθένας παίρνει το δικό του τηλέφωνο γιατί δεν τους καλύπτει η Κομισιόν. Και ε, υπήρχε πρόβλημα επομένω, γιατί ακόμα και για να συνεργαστεί η κυρία Άστον με το Συμβούλιο, τόσο ώστε να μπορέσει να δώσει αυτό το οποίο έπρεπε για να γίνει ταχύ ανάπτυξη. Οπότε συνέχεια έχουμε μια, μια διετία. Μια διετία αφού ε, φτιάξαμε την εξωτερική υπηρεσία, είμαστε σε αυτήν την κατασκευή. Για μένα αυτό είναι ακατανόητο. Πέραν των πολιτικών ζητημάτων, αυτό ε, είναι ένα φρένο όσον αφορά την ε, εύρυθμη ανάπτυξη των αποστολών. Τώρα, για τα, τη διπλωματική πλευρά του πράγματος, ο Ρωμάνο Πρόντι που εδώ το ξέρουμε καλά, ε, διορίστηκε διαμεσολαβητής από πλευράς ε, ΟΗΕ. Τι γίνεται εδώ πέρα λοιπόν, πώς αυτό θα συναρθρωθεί, πώς, πώς θα κολλήσει σε αυτά τις προσπάθειες η, Ευρωπαϊκή Ένωση, στις προσπάθειες λοιπόν του ΟΗΕ και του Πρόντι, βλέπουμε ότι δήλωσε και εμείς κάναμε μια αποστολή ως ΑΦΕΤ ε, στη Νέα Υόρκη και όλοι, όλοι, όλοι στον ΟΗΕ μας είπαν ότι θεωρούσαν ε, ότι με τίποτα δεν γίνεται στρατιωτική επιχείρηση ε, πριν τον Σεπτέμβριο του 2013. Οπότε για άλλη μια φορά είχαμε την εντύπωση ότι έχουμε μείνει πίσω σε σχέση με τον κατεπήγονα δεν δηλαδή τα χαρακτήρα της πραγματικότητας και να δούμε επομένω ακριβώς πώς μπορούμε τελικά εμείς να συνοηθούμε, να συντονιστούμε με τον Ρωμανό Πρόντι για αυτές τις προσπάθειες που καταβάλλονται ή για τις δημοτικές προσπάθειες. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Έχουμε και τον κύριο Παντζέρη για την ε, αντιπροσωπεία των σχέσεων με το Μαγρέπ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ ότι πρέπει να σκεφτούμε τα λάθη μας, ε, τα λάθη κατανόησης κυρίως τα λάθη που κάναμε, γιατί είναι σίγουρο ότι η παρουσία της μαγκρεμπίνικης αλκάιτας είναι συνέπεια των λάθος χειρισμών κατά της τρομοκρατίας που κάναμε μετά την 11η Σεπτεμβρίου και εμείς αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια. Γιατί ένα από τα βασικά θέματα που είναι και οικονομικό θέμα είναι ότι στο νότο της Αλγερίας και στο βόρειο Μαλή εξαφανίστηκε μια βασική πηγή ε, εισοδήματος που, που υπήρχε και ήταν ο τουρισμός. Δεν υπάρχει πια αυτός και αυτό δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στον πληθυσμό. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Το να ερμηνεύσουμε λοιπόν την κρίση του Μαλή ως ε, βασικά έμεση συνέπεια, άμεση συγγνώμη, συνέπεια της λιβικής κρίσης ή της αραβικής άνοιξης δεν είναι απόλυτα σωστό. Γιατί μετά από 20 χρόνια δημοκρατίας εντός εισαγωγικών ε, είχαμε τους τεράστιο πρόβλημα ανάμεσα στο πολιτικό κατεστημένο ας πούμε και στον πληθυσμό στον Παμάκο. Είχαμε απίστευτο μηχανισμό διαφθοράς, ε, η κοινωνία έφτασε στα όρια της ρήξης. Νομίζω ότι για να καταλάβουμε τι γίνεται στο Μαλί, πρέπει να τα συνειδητοποιήσουμε όλα αυτά. Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε το Μαλί, πρέπει να τα συνειδητοποιήσουμε όλα αυτά. Ε, η κοινωνική ανάπτυξη ε, έγινε ουσιαστικά γύρω από την ε, πρωτεύουσα ε, εις βάρος του Βορρά, εις βάρος της υπόλοιπης χώρας. Αυτό είναι σημαντικό να το λάβουμε υπόψη μας. Επίσης υπάρχει μια αντιφαντική κατάσταση και στις ε, όμορες χώρες. Γιατί σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Αλγερία και η Μαυριτανία ενδιαφέρονται ε, δεν θέλουν να ε, προωθηθούν ας πούμε, οι τρομοκρατικέ δράσεις, δεν θέλουν να εξαχθούν οι τρομοκρατικέ δράσεις. Υπάρχει απ' την άλλη ο Ε, που ζει μια τελείως άλλη πραγματικότητα. Τους τελευταίους μήνες έγιναν πολλά πράγματα χωρίς κανένας να παρέμβει σε, στην περιοχή του Νίγηρα. Το θέμα των όμορων χωρών είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό να γίνει μια διπλωματική προσπάθεια και σημαντικό είναι να συμμετάσχει και το Μαρόκο. Τέλος, υπάρχει ένα πολύ λεπτό θέμα της ε, ανεξαρτησίας του, του Αζαουάντα. Θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις διάφορες κινήσεις. Το, Εθνικό Κίνημα Απελευθέρωσης του Αζαουάντα. Ξέρετε, τον, ξέρετε ότι ο, ο αρχηγός έγινε δεκτός πολύ θερμά ε, σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και από κάποια ΜΜΕ ευρωπαϊκά. Ε, δεν νομίζω ότι σήμερα υπάρχει μια ενιαία θεώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Α, ασφάλεια, αποκατάσταση της εδαφικής συνοχής και τρίτον, ε, πολιτική Κοινωνική συνοχή. Δεν, το βλέπουμε, δεν τα βλέπουμε καθόλου με τον ίδιο τρόπο αυτά τα τρία επίπεδα. Νομίζω ότι αφήσαμε τα πράγματα να ξεχαρβαλωθούν επί πάρα πολύ καιρό και προσπαθούμε να επιλύσουμε τώρα την κατάσταση. Ευχαριστώ, ε, τον κύριο Κέρκοφ θέλω να να ρωτήσω ακριβώ πώ επέδρασε στις εξελίξεις στην περιοχή ο θάνατος του Μπιν Λάντεν και η κατάτμιση, η πολυδιάσπαση τέλος πάντων Αλκάιδα. Πώς επέδρασε η, η, η εσωτερική αλλαγή που έγινε στη δομή της Αλκάιδα. Ευχαριστώ κύριε Νικολάγιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η κατάσταση στο Σαχέλ και στο Μαγκρέπ ε, όλο ένα και περισσότερο έχει το χαρακτήρα του κατεπίοντος κατά κάποιο τρόπο γιατί η Αλκάιντα αλλάζει στρατηγική της και έχουμε τώρα κάποια, κάποια κράτη τα οποία είναι αποδιοργανωμένα, ξεχαρβαλωμένα Α, όπως ας πούμε το τι έγινε Έχουμε την άλλη μεριά, έχουμε τη Σενεγάλη, η οποία βέβαια είναι η φωτεινή εξαίρεση, οπότε μπορούμε Μπορούμε να έχουμε τη Σενεγάλη πλέον ως βάση για να δράσουμε. Και τέλος πάντων έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, όσον αφορά το, το, τι έγινε, το, το, τι γίνεται μάλλον στη Λιβύη μετά την ε, πτώση του καθεστώτος ε, ε, Καντάφη. Τώρα θα δούμε κατά πόσο μπορεί το κράτος τώρα να προστατεύσει τον οπλισμό ο οποίος υπάρχει, γιατί έχουν πάρα πολλά ελαφρά όπλα Πάρα πολλά από αυτά τα καταλήγουν στο Σαχέλ. Δεύτερη ερώτηση. Το θέμα είναι το πώ εμείς δυσκολευόμαστε να προσλάβουμε προσωπικό για την αποστολή στον Ήγηρα. Θεωρείτε ότι πρόκειται για κάποια δυσκολία η οποία οφείλεται στο περίπλοκο της διαδικασίας ή μήπως πρόκειται για δυσκολία η οποία έχει συγκυριακό χαρακτήρα. Υπάρχει κάποιο βάση δεδομένων για τους εμπειρογνώμονε μα, οπότε να μπορεί να διερευνηθεί το πρόβλημα, γιατί η, η επέμβαση εκεί και η παρέμβαση τέλο πάντων θα πρέπει να έχει επίγοντα χαρακτήρα. Γιατί άμα αρχίσουμε τις συνομιλίε, τις επαφές, τις διαπραγματεύσει, τότε τα πράγματα θα πάνε στο χειρότερο στην περιοχή. Merci. ευχαριστώ. Η κυρία Κοπά το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούγοντάς σας και μετά από τη συνολική εικόνα που μας έχετε παρουσιάσει για την κατάσταση του Σαχέλ, συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλια βέβαια του Προέδρου του κ. Ντανσόν, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε βαφτίσει ως συνολική αντιμετώπιση για το Σαχέλ έχει αποτελέσει μια πλήρη καταστροφή. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν επέτυχε πουθενά. Δεν έχουμε αποτρέψει την επιδείνωση της κατάστασης στο Σαχέλ. Το να συνεχίσουμε λοιπόν να συζητάμε το θέμα αυτό με την προσέγγιση αυτή σαν να μην συμβαίνει τίποτα δεν νομίζω ότι βοηθάει καθόλου. Φαίνεται αυτή τη στιγμή αδύρυτο ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και υπό, υπό μια στρατιωτική πτυχή, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν συγχρόνως και ειρηνιστικοί ειρηνικέ δράσει παράλληλα. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που θα πρέπει να αναδιαρθρώσουμε τη στρατηγική μας για την περιοχή. Δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Καταρχήν, έχουμε πρόσφατα ενεργοποίησει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρήσεων στο κέρας της Αφρικής. Πιστεύετε ότι αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τις επιχειρήσεις στο Σαχέλ. Μπορείτε να φανταστείτε έναν τρόπο με τον οποίο αυτή η κινητοποίηση του κέντρου επιχειρήσεων μπορεί να παίξει ρόλο για τις τρεις αποστολές στο Σαχέλ και σε σχέση με την περαιτέρω ανάπτυξη της ΚΕΠΑ. Πιστεύετε ότι οι δράσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν ένα υπόδειγμα να χρησιμοποιήσουμε άλλες περιοχές όπως αυτές που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η δεύτερη μου παρατήρηση είναι η εξής βάσει των πληροφοριών που έχουμε, υπάρχει ένας κίνδυνος να υπάρξει διασπορά πυρηνικού υλικού στο Σαχέλ με πολύ σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια ασφάλεια. Μήπως μπορείτε να αναφερθείτε στις ενέργειες που θα κάνει η EU στον Ήγηρα για την ε, ε, ασφάλεια του, των αποθεμάτων ουρανίου στο Βόρειο Νίγηρα. Ο κύριος Κέλαμ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας για την ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου πληροφόρηση που μας έχουν δώσει, αλλά και εγώ τίνω να συμφωνήσω ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σαχέλ δεν έχει επιτύχει ακόμα τους στόχους της. Η κατάσταση λοιπόν είναι ανησυχητικότερη από ό,τι στο παρελθόν. Και το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να σπάσουμε ένα φαύλο κύκλο ε, για να σπάσει αυτή η πολιτική αστάθεια. έχουμε τις εγκληματικές ομάδες, ε, τους μαχητές του Ισλάμ, ε, τον, τους λαθρεμπόρους ναρκωτικών, όλοι αυτοί συγκεντρώνονται και εξαπλώνται στην περιοχή. Συμφωνώ λοιπόν με την κυρία Κοπά ότι μπορεί να γίνει τελικά ένα παγκόσμιο πρόβλημα που να οδηγήσει σε παγκόσμια αστάθεια. Επομένως η αντίδρασή μας σε αυτό είναι πολύ σημαντική. Ένα σημαντικό μήνυμα, θετικό μήνυμα, είναι ότι τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να συμφωνήσει για επιπλέον ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, μην ξεχνάτε ότι 200.000 παιδιά πεθαίνουν σε αυτή την περιοχή κάθε χρόνο. Αυτό είναι το background. Το θέμα είναι αυτή τη βοήθεια πώς θα την ε, καναλιζάρουμε, πώς θα την δώσουμε στον πληθυσμό χωρίς διαμεσολάβηση, χωρίς διαμεσολαβητές. Ένα ενδιαφέρον σχόλιο ακούστηκε από τον κύριο Λόπες Μπλάνκο ότι ακόμα και η περίπτωση διεθνούς παρέμβασης μπορεί να οδηγήσει σε συμμαχίες διαφόρων ομάδων ε, ή μάλλον να τις αναγκάσει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, αν δεν έχουμε μία παράλληλη ε, πολιτική λύση πέρα από τη στρατιωτική αποκλείεται αυτή η διεθνής παρέμβαση να έχει επιτυχία. Η περιφερειακή συνεργασία είναι πολύ σημαντική. Είναι πιο αδύναμη από ό,τι θα μπορούσε να είναι και συμφωνώ με την ιδέα σας ότι η Αλγερία θα πρέπει να εμπλακεί τις προσπάθειές μας. Το ανησυχητικό είναι αυτά που είπε ο συνάδελφος στην έκθεσή του ότι σκοντάφτη η ευρωπαϊκή αποστολή, η ευρωπαϊκή επιχείρηση, δεν είναι ακόμα πλήρως επιχειρησιακή, ε, που σκοντάφτει σε γραφειοκρατικά εμπόδια. Οι συνεντεύξεις με το προσωπικό, η εξεύρεση πόρων για να ξεκινήσει αυτά είναι εμπόδια ανησυχητικά. Χρειαζόμαστε καλύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Τελευταίο ερώτημα έχοντας υπόψη το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. όπου προτείνεται πάγωμα του προπολογισμού ή ίσως και περικοπές του. Πώς βλέπετε τις προοπτικές να βρούμε τα απαραίτητα χρήματα για βοήθεια σε αυτή την περιοχή, η οποία περιοχή χρειάζεται μεγαλύτερη βοήθεια, υπό διαφορετικές μορφές. Πώς ε, δικαιολογείται η περικοπή τη στιγμή που χρειάζομαστε περισσότερα λεφτά για αυτή την πολιτική. Ε, ο κύριος Κέρκοπ το είπε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα από αυτά που κάναμε μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ. Η Άννα Γκόμες, τελευταία ομιλήτρια. Συμφωνώ 100% πρόεδρε με τα όσα είπε ο κ. Ναι, ναι, θεωρώ ότι είχαμε χαθεί πάρα πολλοί χρόνος. Και οι συνέπειε τη κρίση στην Ευρώπη δεν είναι μόνο οικονομικού χαρακτήρα, είναι και πολιτικού χαρακτήρα και ακριβώ έτσι εξηγείται το ότι με δεδομένου αυτού όλου του κινδύνου που όλοι έχουν διαπιστώσει ότι σοβούν τόσο πολύ καιρό, δεν έγινε τίποτα. Και ακόμα αυτά τα οποία κάνουμε, τα κάνουμε τόσο, τόσο, τόσο αργά και, και με τόσα προβλήματα τι θα γίνει, δεν υπάρχει κάποιο είδους αποθεματικό. Για πέστε μου τι γίνεται με, με αυτό το θέμα, γιατί να καταλάβω επίση, για πέστε μας τι γίνεται από πλευρά τη συμβολή των κάτω γιατί α, βλέπω με τι γίνεται στη χώρα μου. Θα έπρεπε, θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Καλά, είναι τώρα, έτσι, λόγω τη οικονομική συγκυρία δεν μπορούμε να, να βοηθήσουμε, αλλά τέλο έχουμε ένα σωρό κόσμο ο οποίο ε, ξέρει, ξέρει το θέμα και θα μπορούσαν αυτοί να βοηθήσουν ε, μετά. Επίση έχουμε το θέμα τη Λιβύη και το πώ και εκεί έχουμε χάσει. Έχουμε τόσο διασπαθήσει πόρους. ανοίξαμε και την υπηρεσία μας, τη Βαγκάζη, οπότε μετά τίποτα. Μετά, φτιάξε, μετά στείλαμε άλλη αποστολή στην Τρίπολη. Επομένως, τίποτα δεν κάναμε με όλα αυτά τα οποία γνωρίζαμε ότι εκεί είναι δεδομένα και θα έπρεπε να είναι χρήσιμα για όλους την περιοχή. Πήγα στο Ζιντάν πρόσφατα, εκεί έξω από την Τρίπολη Και πήγα και πέρα σε κάποια μεγάλη πυρτίδα αποθήκη, τέλος πάντων αποθήκη πυρομαχικών που υπήρχε από την εποχή του Καντάφη. Τώρα έχουμε 72 υπόστεγα μεγάλα γεμάτα με όπλα. Εντάξει, θα τα φυλάει το ΝΑΤΟ, αλλά άμα πέσει και καμία βόμβα, φαντάζεται τι θα γίνει. Είναι όλα αυτά τα αυτή τη τεράστια έκταση τέλος πάντων <clears throat> γεμάτη με βόμβες, όπλα κλπ. Α, δεν μπορούσα να, φέρω και μαζί για να σας το δείξω, αλλά τέλος πάντων και υπάρχει εκεί πέρα η μη κυβερνητική οργάνωση που δουλεύει, αλλά δεν έχουν, δεν έχουν αυτά που χρειάζονται. Και θεωρούν ότι θα μπορέσουν τελικά σε έξι χρόνια να δημιουργήσουν συνθήκες ασφαλείας για αυτές τις εγκαταστάσεις. Και ξέρετε, η Λιβύη είναι γεμάτη με τέτοιες εγκαταστάσεις αυτή που σας περιέγραψα. Άρα, άρα είναι προφανές ότι θα πρέπει να κάνουμε πολύ πολύ περισσότερα. Και μην μου λέτε ότι εκεί πέρα δεν υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει χάος και τώρα μπορούμε να βοηθήσουμε την νέα κυβέρνηση. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Πήγα εκεί, μίλησα με ναι, τι τοπικέ αρχέ του Ζιντάν που μα ζήτησαν να πάμε να του δούμε και μα είπαν τι γίνεται, βοηθήστε μα, δεν κάνετε τίποτα γιατί βλέπουν ότι υπάρχει κίνδυνος για τους ανθρώπους τους και έχουμε εκεί πέρα ένα σωρό με οργανώσει και είναι δύο Ολλανδοί, διάφοροι ξένοι. Μη μου λέτε ότι <clears throat> δεν υπάρχουν συνθήκε και προποθέσει για να αρχίσουμε να, <clears throat> συγγνώμη, να δουλεύουμε στη Λιβύη. Να, τι γίνεται με τα προβλήματα αυτά. Επίσης, Έχουμε ένα σωρό άλλα θετικά για τη Λιβύη. Έχουμε την τρομοκρατική επίθεση κατά του Αμερικανού πρέσβη και του προσωπικού. Ήταν τρομερή αντίδραση του πληθυσμού. Γιατί ουσιαστικά αυτοί αποθήσανε τους τρομοκράτες. Σηκώθηκαν και φύγανε από την Πενγκάζη. Και πήγαν κάπου αλλού βέβαια στη Λιβύη και χρησιμοποιούν ε, αυτές τις περιοχές που δεν τις ελέγχει κανείς για να κάνουν τη δουλειά του. Τέλο πάντων θα πρέπει να χαραχτεί κάποια στατική, θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερο. Επίση, είναι και το θέμα της Σαχάρας. Και θυμάμαι το 2004 είχα πάει στο Τιντούφ και είχα γράψει και ένα άρθρο και έλεγα ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ είναι πλέον όριμοι να στατολογηθούν από του Τρομοκράτε. Είχαν παράπονα στη Σαχάρα επιβάλλεται να υιοθετήσουμε κοινή θέση που δεν έχουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα θα πρέπει εκεί να βάλουν τα πράγματα σε κάποια σειρά. Τι γίνεται και με το Μαρόκο. Να, επομένω, από πού αντλούν κόσμο τρομοκράτε. Γουινία Μπισάου. Κύριε Κέρχοβε. Ναι, είναι τρομερό αυτό το οποίο έγινε με τις υπηρεσίες μας που αποχώρησαν. Είχαμε μία αποστολή ε, της ΚΕΠΑ εκεί πέρα. Ε, υποτίθεται ότι έπρεπε να εκπαιδεύσουμε τους ε, στρατιωτικούς, τίποτα δεν είναι, έγινε σωστά η δουλειά, δεν επανδρώθηκε σωστά. Και με το που έγινε το πραξικόπημα, ήταν και το θέμα των ναρκωτικών και εμεί το θεωρήσαμε αυτό πρόφαση για να αποσύρουμε την αποστολή μα. Ε, πώς να μην γίνει τώρα η πέρα του εμπορίου ναρκωτικών. Ε, βέβαια, ήταν βέβαια θα γίνει κάτι τέτοιο. Και υπάρχουν και χειρότερα ακόμα. Ποιο βρίσκεται πίσω από το πραξικόπημα αυτό, που φυσικά το πραξικόπημα βοηθάει τους ε, του εμπόρους ναρκωτικών, το ΣΕΝΤΕΟ, που ήταν υποτίθεται η, η σύμμαχή μας. Και τώρα αντί λοιπόν να τους ε, πολεμήσουν, τους βοηθάνε. Αυτοί ήταν οι συνομιλητές μας. Μήπως θα πρέπει να φροντίσουμε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να συνομιλούμε κάποιον, αλλά Μήπως θα πρέπει αυτό το προβληματάκι να το ρυθμίσουμε. Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για, τον, για, για τους Βαχαμπίτες που είπατε ότι εξαπλώνονται και ε, ενισχύονται στην περιοχή. Πώς θα μπορούσαμε να δούμε τι θα γίνει. γιατί το θέμα εδώ δεν είναι ιδεολογικό, είναι οικονομικό, το ξέρουμε. Και πίσω από αυτούς βρίσκεται η Σαουδική Αραβία. Οπότε γι' αυτό θα ήθελα να, να δω πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια των θεμάτων που θέλουμε, θέλουμε, θέλουμε να μας απασχολήσουν στα πλαίσια αυτών των αποστολών για την ασφάλεια του Σαχέλ. Ευχαριστώ. Εγώ σας προτείνω να δώσουμε το λόγο στους τρεις προσκεκλημένους μας με την σειρά που ακολουθήσανε στις αρχικές παρεμβάσεις και να απαντήσουν στα ερωτήματα που θεωρούν ότι εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους και αν θεωρούν ότι μπορούν να δώσουν στοιχεία απαντήσεως και εάν θέλουν να εκφράσουν άποψη και σε θέματα που δεν τους αφορούν άμεσα και αυτό γίνεται. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν το λόγο. Όλα αυτά τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν και με την χρησιμότητα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να επανέλθουμε και στη λογική και στη φύση αυτής της στρατηγικής και στις προσδοκίες οι οποίες μπορούν να προκύψουν σε σχέση με τα δυνητικά αποτελέσματα. Η στρατηγή του Σαχέλ είναι μια στρατηγή συμβολής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι υποκατάστασης. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα των άλλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιλύσει προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες του Σαχέλ, της Σαχάρας, της Βόρειας Αφρικής. Μόνο μπορεί να βοηθήσει τα κράτη αυτά να αναπτύξουν τις δικές στρατηγικές. Δεν μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε την κυβέρνηση του Μαλή, η οποία καταραίει. Δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε την κυβέρνηση αυτή. Μόνο μπορούμε να βοηθήσουμε να αναδημιουργηθεί η κυβέρνηση αυτή. Και συγχρόνως δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το στρατό του Μαλή ο οποίος είναι διαλυμένος και κατεστραμμένος. Μόνο μπορούμε να βοηθήσουμε <clears throat> να αναδημιουργηθεί αλλά για να υπάρξει μια στρατιωτική δύναμη η οποία βρίσκεται κάτω από πολιτική εξουσία πρέπει να αναδημιουργήσουμε και την ίδια την πολιτική εξουσία. Τα προβλήματα είναι πιο σοβαρά, πιο βαθιά, πιο διαρθωτικά. Μια στρατηγική λοιπόν που έχουμε εγκρίνει πριν από 1,5 χρόνο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχει το θέμα της διαχείρισης των προσδοκιών. Πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι και τα όρια της διεθνούς δράσης. Μπορούμε να ρωτήσουμε γιατί οι ΗΠΑ δεν έχουν λύσει το πρόβλημα. Γιατί οι Κινέζοι δεν έχουν λύσει το πρόβλημα του Σαχέλ. Γιατί όχι η Γαλλία, γιατί όχι το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν στη διάθεσή τους πολλά μέσα. Γιατί η Αλγερία που έχει ένα στρατό πάνω από 300.000 στρατιώτες και η οποία παίρνει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία έχει πολύ μεγάλες υπηρεσίες μυστικές και γνωρίζει πολύ καλά το έδαφος και την περιοχή, γιατί δεν βοηθάει να ανασυγκροτηθεί το κράτος του Μαλή. Γιατί κανονικά θα πρέπει να ήταν ο πρώτος ε, ε, ενδιαφερόμενος για τη σταθερότητα και όχι την αστάθεια του Μαλή. Τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά, πολύ διαρθρωτικά. Το Μαλλί έχει αποαπικιοποιηθεί εδώ και περίπου 60 χρόνια. Βρίσκεται σε ένα επίπεδο ανάπτυξης, σε ένα ιστορικό επίπεδο, όπου τα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δημιουργία ενός εθνικού κράτους δεν έχουν αντιμετωπιστεί πλήρως, όπου υπάρχει όπου η σχέση μεταξύ του κράτους και του συνόλου <clears throat> των πολιτών, το λεγόμενο κοινωνικό συμβόλαιο, και <clears throat> η σχέση της κεντρικής κυβέρνησης με περιφερειακούς, περιφερειακούς πληθυσμούς δεν έχει επιληθεί. Το θέμα του κράτους έθνους δεν έχει επιληθεί. Η δημοκρατία η οποία υπάρχει εκεί ήταν αυτή η οποία μπορούσε να είναι εφικτή τότε που πήρε την ανεξαρτησία το Μάλι. Τώρα πια όμως έχει επιδεινωθεί η κατάσταση και είναι μονάχα μία πρόσωψη αυτή η δημοκρατία. Νομίζω ότι η κρίση της Λιβύης δεν ήταν η, η αιτία της κρίσης στο Μαλί. Ήταν η αφορμή ίσως, αλλά όχι η αιτία. Η αιτία είναι τα εσωτερικά προβλήματα του Μαλί και υπάρχει ένα πρόβλημα λειτουργίας της Αλκάιδα σε ευρύτερο επίπεδο. Στο Μαλί είτε στο Ισλαμικό ε, Μαγρέ που είναι ουσιαστικά μια, ένα εξαγώγημο προϊόν της Αλγερίας. Το Μαλή έχει αντιμετωπιστεί εδώ και πάρα πολύ ε, χρόνο αυτήν την ομάδα σαν κάτι που δεν το ενδιέφερε. Ήταν μια ομάδα Αλγερινών οι οποίοι διέφευγαν από την πίεση των δυνάμεων ασφαλείας της Αλγερίας. Για πάρα πολύ καιρό ο πρόεδρος του Μαλή, ο οποίος τώρα αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα και είμαστε σίγουροι ότι και αυτός έχει μια ευθύνη για τα θέματα αυτά, ζήτησε από τους Αλγερινούς να αντιμετωπίσουν <clears throat> την Αλκάιντα στο Μαγκρέπ, κάτι το οποίο φυσικά δεν έκαναν. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό, όχι ότι θέλουν να υποστηρίξουν τη στρατηγική <clears throat> της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σαχέλ έναντι όλων των επικρίσεων, γιατί είναι γεγονός ότι υπήρξε μια κάποια επανάληψη στα θέματα αυτά και μια κάποια μικρή πρόοδος. Αλλά όλα αυτά βρίσκονται στη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε μια ε, ένωση όπου τα πράγματα γίνονται διαδοχικά και με βελτιώσεις σε κάθε καμπή του δρόμου. Είναι, αν θέλετε, μέσα στη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι στο οποίο εγώ μπορώ να επιμείνω ακόμα είναι ότι θα πρέπει και με το Συμβούλιο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι σημαντικός παίκτη στα θέματα αυτά θα πρέπει να είμαστε σε στενή επαφή. Γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της κοινή της μικτής ε, της ομέρους μάλλον συνέλευσης ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε να υπάρξει αυτή η αποστολή στο Μαλί. Και πήγε ακόμα και στο Μπαμάκο για να πείσει το κοινοβούλιο του Μαλί να κάνει τι απαραίτητε ενέργειε. Όλε οι προσπάθειε είναι απαραίτητε. Για να μιλήσουμε για το Ρωμάνο, <clears throat> πρώτη. Είμαστε σε άμεση επαφή μαζί του και μαζί με την ομάδα του, η οποία ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί πλήρως. Και είμαστε επίσης σε επαφή με τον Σαϊτζινίτ, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Ban moon για τη Δυτική Αφρική και ο οποίος συνεργάζεται με τον Πρόντι. Αλλά ο Ρωμανοπρόντι ακόμα προσπαθεί να κατανοήσει πλήρως ποια είναι η κατάσταση στο Σαχέλ. Αυτό χρειάζεται χρόνο. Ορισμένοι από εσάς γνωρίζετε το Σαχέλ εδώ και μήνες, εδώ και χρόνια, αλλά δεν είναι εύκολο να βρούμε κάποιον ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση στο Σαχέλ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, αν εξαιρέσουμε το Ζιλ βέβαια, αλλά ο Ζήλ έχει πολύ βαθιές γνώσεις για το θέμα αυτό. Είμαστε όμως σε επαφή με τον κύριο Πρόντι. Έχουμε προσκληθεί από τον κύριο Πρόντι για να πάμε σε συνεδριάσεις που προβλέπει να διοργανώσει. Και ο στόχος μας είναι να το βοηθήσουμε όσο είναι δυνατό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι κάποιο με το πολιτικό βάρος του Ρωμάνου Πρόντι μπορεί να παίξει ένα θεμελιώδη ρόλο σε πολλά επίπεδα. Καταρχήν, μπορεί να συγκεντρώσει τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για να ασκήσουν πίεση στον Παμάκο. Σας είπα ότι το πρόβλημα ήταν ότι η διαδικασία θεσμικής μεταρρυθμίσεως στο Παμάκο ήταν βραδία και έχει πια τροχοπεδεθεί σχεδόν πλήρως. Πρέπει εκεί η διεθνής κοινότητα να ασκήσει πίεση. Και θα έχει φυσικά την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τούτο. Μπορεί επίσης να παίξει ρόλο στη διαμεσολάβηση με τις ομάδες του Βορείου Μαλή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε το Ρωμάνο με τις συμπληρωματικές προσπάθειες διαμεσολάβησης, αλλά αφήναντάς του το ρόλο που έχει αναλάβει μαζί με την Μπουρκίνα Φάσο και την Αλγερία για να εξασφαλίσει ότι θα έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όλοι οι εμπλεκόμενοι. Αυτά τα λοιπόν τα σχόλια που ήθελα να σας αφήσω σε αυτό το στάδιο. Δεν θέλησα να σχολιάσω τη Λιβύη. Γιατί δεν νομίζω ότι έχω τις απαραίτητες γνώσεις για κάτι τέτοιο. Και ίσως μπορεί να σας πω βλακίες και δεν αξίζει τον κόπο λοιπόν να το πράξω αυτό. Μια τελευταία παρατήρηση αν θέλετε. για την ε, ε επιχείρηση η οποία είναι υπό προετοιμασία. η επιχείρηση αυτή, ακόμα και αν φαίνεται καταρχήν ότι η κατάρτιση είναι κάτι εκτός εορτής ή δεν έχει ιδιαίτερο νόημα για την επίλυση του προβλήματος, για μένα είναι η καρδιά της λύσης του προβλήματος. Γιατί τα προβλήματα της αστάθειας στον Παμάκο είναι το αποτέλεσμα ενός στρατού ο οποίος έχει κατακαιρματιστεί, έχει διαλυθεί και ο οποίος ασκεί την πολιτική εξουσία ουσιαστικά. Είναι ένας στρατός που δεν έχει πια λυσίδα ε, εξουσίας και ιεραρχίας και όπου οι λοχίες δίνουν διαταγές στους στρατηγούς. Πρέπει λοιπόν να αναδημιουργηθεί ένας πραγματικός στρατός για το Μαλί που να έχει μια ιεραρχία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζει ο Οργανισμός των Εθνών. Είναι απαραίτητο για να μπορέσει να λειτουργήσει το πολιτικό σύστημα στο Μαλί. Μια άλλη πτυχή είναι ότι η επαναφορά της ιεραρχίας και η επαναφορά των λειτουργικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων του στρατού του Μαλή και αυτό περιλαμβάνει και την ε, κατάρτιση για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την προστασία των αμάχων. Αυτό είναι το κλειδί για την αξιόπιστη χρήση της βίας που θα οδηγήσει όλους τους εμπλεκόμενους στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει και τη διεθνή κοινότητα. Η, δράση αυτή που γίνεται από τη φύσμα δεν έχει σε στόχο να κάνει πόλεμο στον Βορρά. Είναι απλώς σε υποστήριξη του στρατού του Μαλή και που θα συνοδεύσει μια προσπάθεια διαπραγματεύσεων με τις ε, ομάδες του Βορρά και ιδίω με τον πληθυσμό του Βορρά, γιατί αυτοί θα έρθουν στο τραπέζι. Οι υπεύθυνοι λοιπόν σε επίπεδο κοινότητος και σε επίπεδο φυλών, αυτοί θα πρέπει να εμπλεκούν και όχι μονάχα οι επικεφαλής των ε, ανταρτών εκεί. Για να υπάρξει όμως μια δυνατότητα άσκηση πίεση από την κυβέρνηση του Μαλή, θα πρέπει να έχει μια ελαχίστως επαρκή στρατιωτική δύναμη με την υποστήριξη του διεθνού κοινότητα. Εμεί σα ευχαριστούμε που μα ε, εξηγήσατε τι εξελίξει και τώρα έδινε τον κύριο Χάμπερ. Κύριε Πρόεδρε, οι ερωτήσει που μου υποβλήθηκαν είναι ερωτήσει που ξεπερνούν τα θέματα τα οποία τώρα συζητούμε αυτέ τι αποστολέ. γιατί οι ερωτήσει ήταν οριζόντιου χαρακτήρα οπότε χρειάζομαι κάποιο χρόνο για να σα τα εξηγήσω ε, εγώ ευχαρίστω. Ε, Πώ σα εξαρτάται. Εντάξει, πολύ καλά. Το θέμα δεν είναι τα χρήματα. Αυτά είναι τα καλά νέα. Η, ο, η πρικοδότηση τέλο πάντων τη ΚΕΠΑ αρκεί για όλε τι αποστολέ μα και ακόμα και σε σχέση με την ε, προβολή του, μεσοπρόθεσμου προπολογισμού θα έχουμε περίπου 360 εκατομμύρια το χρόνο που φτάνουν και περισσεύουν για τις αποστολές αυτές γιατί θα πρέπει να απορροφήσουμε να χρησιμοποιήσουμε 200. Το υπόλοιπο είναι ελεγκτικά μέτρα, τέλος πάντων, άλλα πέρα των αποστολών. Επομένως, το θέμα δεν είναι το αν λεφτά υπάρχουν, είναι η δυσκολία του να εκταμιαυτούν αυτά τα χρήματα. Άλλο πρόβλημα, το προσωπικό. Και αυτό καταρχήν είναι πρόβλημα. Γιατί, γιατί καταρχήν έχουμε ένα φυσικό όριο 4.000 από αποσπάσεις, από προσλήψεις τοπικών και μη. Αυτό θέλω να μας δώσουν σαν ανθρώπινους πόρους τα κράτη-μέλη. Όμως, όμως, φέτος έχουμε 200 λιγότερους από πέρσι. Όμως έχουμε τρεις αποστολές παραπάνω. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί λόγω του κοσυφοπεδίου τόσο, γι' αυτό συνεχιστεί το Κόσοβο τροφοδοτούσε τις άλλες αποστολές από προσωπικού. Οπότε τώρα θα προωθήσουμε λιγότερα χρήματα για το ίδιο πλαίσιο. Το πρόβλημα με το προσωπικό είναι το εξής. Έχουμε για κάθε θέση 1,7 υποψηφίους. Καταρχήν αυτό φαίνεται αρκετό αλλά δεν είναι. Γιατί όλοι θέλουν την ίδια θέση και δεν πάνε στις άλλες θέσει. Δεν ενδιαφέρονται. Οπότε πρέπει να βρεθούμε στα κράτη-μέλη και να τους ζητήσουμε να προσλάβουν προσωπικό και όχι να αποσπούν οι υπαλλήλου. Οπότε και αυτό είναι η διαδικασία χρονοβόρα. Θα λυνόταν το πρόβλημα αν μπορούσαμε να προσλάβουμε. Αλλά τα κράτη-μέλη για οικονομικού λόγους επιμένουν στη μέθοδο της απόσπασης. Αν τώρα υπολογίσετε τη συμβολή από πλευράς αστυνομικών, στρατιωτικών κλπ. Ανά εκατομμύριο κατοίκων έχουμε μέχρι και 100 μονάδες απόκληση μεταξύ του, του, του, του καλύτερου και του χειρότερου. Επομένως. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχει ανισομέρειο όσον αφορά τις υποχρεώσεις. Και καταρχήν έχουμε προσωπικό για να επανδώσουμε τι αποστολέ. Καταρχήν. Τώρα, εάν μου πείτε ποια είναι η βασική αιτία των καθυστερήσεων για φέτος. Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι η απουσία βαστικών μέτρων που ξέρετε έχουμε αυτές τις τρεις νέες αποστολές και ετοιμάζεται και άλλη μία στην Λιβύη. Θα ανασκοτήσουμε την Γιούμπεν Ράφα και από πλευράς προγραμματισμού έχουμε την πολυεπίπεδη άσκηση. Αυτό ήταν γυμνάσιο, τέλο πάντων άσκηση επί χάρτου και όχι πραγματική αποστολή. Αλλά έτσι όμως, έτσι φτάσαμε στα όρια των δυνατοτήτων μας και των πόρων που έχουμε. Αυτά όσον αφορά τις επίσης. Τώρα, επιτόπου όταν πήγα στην Γεωργία προ τέτρα τετραετίας, υπήρχε εκεί προπαρασκευαστικό μέτρο προπαρασκευή τέλο πάντων. 6 Αυγούστου και 6 Σεπτεμβρίου υπήρχαν κάποιες ρυθμίσεις και ταυτόχρονα έγιναν τα προπαρασκευαστικά μέτρα. Σεπτέμβριο αποφάσισε το Συμβούλιο, 21 Δεκεμβρίου προσλήφθηκα και έπρεπε τότε να... Αν έπρεπε λοιπόν τότε να αρχίσω εγώ να, να, να, να βρίσκω το, εγκαταστάσει, τηλέφωνα κλπ. Ποτέ θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτά τα οποία κάναμε και αποφασίσαμε να γίνουμε στη Γεωργία από την 1η Οκτωβρίου. Οπότε βεβαίω και ε, ήταν γρήγορη, σύντομη διαδικασία προσκευή, αλλά πολύ αποτελεσματική. Είχαμε τέλο και προσωπικό. τώρα για το κόσμο Εκεί δεν είχαμε προπαρασκευαστικά μέτρα με την καθαρή έννοια, αλλά υπήρχε κάποια αποστολή που έγινε αμέσω μόλι αγγελήθηκε η ανεξαρτησία. Είχαμε επομένω το, το, το, το, πρόγραμμα Χτισάρι, πήγε ένα χρόνο να προετοιμάζω και υπήρχαν επομένω τα προπαρασκευαστικά μέτρα. Όμω τίποτα από αυτά δεν ίσχυσε για τι νέε αποστολέ. Γι' αυτό ακριβώ και μιλούμε περί καθυστέρηση. Και δεν είναι ο Νίγερ χειρότερη περίπτωση. Η Σομαλία. Η Σομαλία να δείτε τι γίνεται. Υπάρχουν και διάφοροι παράγοντε εκτό ελέγχου. Και δεν κάνει και θέμα η απουσία προπαρασκευή. Τώρα, τα καλά νέα είναι ότι στο μεταξύ συμφώνησε η Επιτροπή να γίνουν μέτρα προπαρασκευή για τι νέε αποστολέ. Οπότε, ή στο μέλλον θα μας ωφελήσει αυτή η απόφαση. Πάντως προς το παρόν δεν κάνει διαφορά. Δεν βοηθάει τι αποστολέ. Ούτε την Ιούμπαν Ράφα, διότι η ίδια αυτή η αποστολή έχει αναπτυχθεί. Αυτά. Καταρχήν τώρα το άλλο θέμα είναι το εξή. Για αυτές τις αποθήκες. Το υλικό θα βγει από τις αποθήκες μας που ήδη έχουμε ας πούμε στη Βοσνία Ζεγοβίνη Εκεί έγιναν μεγάλες περικοπές στο υλικό, οπότε υπάρχει υλικό. από εκεί. για το UCAP, εκεί είναι μια μεγάλη πρόκληση, διότι στην αποστολή UCAP εκεί έπρεπε να γίνουν συμβάσεις για μια εταιρεία επιμελητίας για να μπορέσουμε να έχουμε ό,τι χρειαζόμασταν και αυτό συνεπεί για το καθυστέρηση έξι εβδομάδων για να γίνει αυτός ο διαγωνισμός. Διότι έπρεπε να να γίνουν τα πράγματα όπως προβλέπονται από τον κανονισμό. Και ο κεφαλή αποστολής ακόμα περιμένει να έρθουν τα, αυτοκίνητα, να έρθουν ό,τι, ό,τι πρέπει τέλο πάντων να έρθει από τη Βοσνία. Αλλά στο βάθος του τούνελ υπάρχει φως. Άλλο πρόβλημα. Όπως γνωρίζετε. Ε, νομικά τα πάντα για την αποστολή εξαρτώνται από τον επικεφαλής πάει η Κομισιόν, βάζει το λογαριασμό 25 εκατομμύρια και αυτός μετά κανονίζει. Αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Και άλλα προβλήματα όσον αφορά το προσωπικό. Δεν, δεν ισχύει για, τους, ε, για όσους υπηρετούν τις αποστελές αυτές ό,τι ισχύει για τους υπαλλήλους εδώ στις Βρυξέλλες. Πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό, το FBI και με, με άλλους συναρμόδιους διευθυντές στην Επιτροπή γίνονται επαφές, βρίσκονται εξελίξει, αλλά συνεχίζονται. Και εν πάση κάθε νέα αποστολή πρέπει να ξεκινάει από το 0, από το α. Και αυτό είναι καθυστέρηση. Και σε κάθε χώρα υπάρχει διαφορετικό σύστημα, η διαφορετικό σύστημα έχει κάθε αποστολή. Οπότε κάθε φορά ξεκινάμε από το α. Αυτά έχουμε και τα καλά και τα κακά νέα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο, αλλά κατά κάποιο τρόπο με αυτές τις τρεις αποστολές ε, ε, κατά κάποιο τρόπο βιαστήκαμε σε ένα χρόνο αν γινόντουσαν θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Αυτό θέλω να σας πω, ότι δεν πρόκειται για δική μας έλλειψη προσπάθειας. Απλώς είναι συγκυριακές οι αιτίες του προβλήματος. Και από ένα συγκεκριμένο σημείο και μετά εμείς ε, παίρνουμε τη σκητάλη και είμαστε αρμόδιοι γιατί μέχρι ένα σημείο όλα αυτά από τα κράτη-μέλη. Να, στη Σομαλία τι έγινε. Επί δύο χρόνια προσπαθούσαν να τα βρουν τα κράτη-μέλη μέχρι όταν εγκριθεί η αποστολή. Προέτους δηλαδή. από εκείνο το σημείο και μετά, όντω εμεί έχουμε την αρμοδιότητα και την ευθύνη και την αποδεχόμαστε. Και έχουμε τι συνθήκε που έχουμε για να δουλέψουμε. Αλλά πριν, πριν από αυτό το χρονικό σημείο, τα κράτη-μέλη έχουν την ευθύνη και οπότε σε αυτούς να τα πείτε. Τώρα το κέντρο των επιχειρήσεων. Πολιτικό σύμβασμό. Από κρατών μελών δεν μπορούσε να κάνει μία αποστολή με υποστηρίζει και με ευγνώμων, αλλά, αλλά στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα και με, με, με 16 υπαλλήλου που έχει το κέντρο επιχείρησεων, δεν μπορούσα να κάνω και πολλά περισσότερα. Ουράνιο και Βόρειο Μαλί. Καταρχήν, καταρχήν θέλαμε να υπάρχει μια υπηρεσία στην, στο Βόρειο Νίγηρα, αλλά μετά για λόγους ασφαλείας το μετανιώσαμε γιατί ε, έχουμε στο ε, νου για το τι πρέπει να κάνουμε με την ε, Λιβύη και όπως θυμάται και ο Μανουέλ τελικά το κράτος υποδοχής οφείλει κάτι να κάνει και θα πρέπει οριζόντια να, να, να προχωρήσουν πριν κοιτάξουν το θέμα της ασφαλείας. Και αυτό είναι γενικότερο θέμα. Τα κράτη υποδοχής συνήθως είναι σε πολύ καλύτερη ε, κατάσταση, πολύ, πολύ μεγάλε δυνατότητε να ελέγξουν τα πράγματα επί τόπου. Να, στο Κόσοβο. Η καταπολέμηση εκεί τη διαφθορά εμποδίζεται από το ότι δεν ομιλούμε τη γλώσσα, <coughs> δεν γνωρίζουμε την νοοτροπία και ο κάθε Κωσοβάρος ξέρει πολύ περισσότερο από όσα η αποστολή. Άρα θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε, θα πρέπει να, να, να ξυπνήσουμε να κάνουμε τόσο πάντων πιο επαγγελματική την αστυνομία του κάθε τόπου. Να, να γιατί. Να, γιατί σηκωθήκαμε και φύγαμε από την Βουενέα ε, Μπισάου και θα πρέπει να αποδεχθούμε το ότι δεν μπορεί να πετυχαίνει κάθε αποστολή. Κάθε φορά είναι, πρόκειται για άλμα στο κενό. Και Κάθε φορά, εν πάση αν δεν έχουμε τι συνένεση και σύμφωνη γνώμη του, του, του, τη τοπική κυβέρνηση, δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό και έχουμε και αυτή την ε, διευθυντική αποστολή στην Τρίπολη και τα πρώτα μαντάτα είναι καλά. Έχουμε έτσι επαφή με όλου, αλλά είναι θέμα τι θα κάνουμε με την ασφάλεια, μια που δεν ε, ε ξέρουμε ακριβώς τι, τι, τι, τι ισχύει στην περιοχή, δεν είμαστε εξοικειωμένοι και φυσικά έχουμε και αυτό το, το καθήκον να τους εξυπηρετήσουμε. Δεν μπορούμε αυτό να το ξεχάσουμε. Αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Να προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα που δεν απαντήσαν οι συνάδελφοι. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι για τα χρονοδιαγράμματα και τις υποθεσμίες. Όντως έπρεπε να είχαμε παρέμβει πολύ νωρίτερα. Αλλά αυτό ήταν βασικά πολιτικό θέμα, δεν υπήρχε συνένεση σε πολιτικό επίπεδο. Πέρα από τις διάφορες ε, δυσκολίες που ανέφερε ο συνάδελφος, αν πάρουμε την περίπτωση του Νίγηρα και τη θεσμική κατανομή αρμοδιοτήτων. Το UCAP Νίγηρας ε, το είχε η, Ευρω... η εξωτερική υπηρεσία η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης. Ενώ το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της δημοκρατίας ήταν ευθύνη της Κομισιόν. Υπάρχει και κατανομή αρμοδιοτήτων. Επίσης, συμφωνώ με αυτό που είπε ο Μανιουέλ για τις βαθιές αιτίες της κρίσης στο Μαλί. Ε, συμφωνώ επίσης ότι ήταν μια επιφανειακή δημοκρατία ε, διαβρωμένη από τη διαφθορά και η Λιβύη ήταν απλώς η αφορμή, ο καταλήτης και όχι η βαθιά αιτία. Ε, για αυτά που υπόθηκαν για τον Ήγηρα. Δεν είμαι πολύ ειδικό για τον Ήγηρα, αλλά είμαστε εντυπωσιασμένοι από, τις, από τη συνοχή των πολιτικών, των αναπτυξιακών πολιτικών για τον Ήγηρα. Ε, και εδώ πέρα νομίζω ότι έχουμε παρέμβει πολύ νωρίτερα από ό,τι στο Μαλί και υπάρχει θέληση να βρούμε ε, συμβιβασμό με τις διάφορες εθνοτικές ομάδες, ε, με τους του και τα λοιπά. Και πρέπει να τις υποστηρίξουμε διάφορα εργαλεία και δεν είμαι τόσο αρνητική όσο εσείς για τον Ήγηρα. πρέπει να εμπλέξουμε το Μαρόκο και την Αλγερία. Φυσικά ήμουνα στο Μαρόκο για την, το θέμα της ομοκρατίας και για το Σακέλ και στο Μαρόκο εξεπλάγην από τις πολλές πληροφορίες που έχουν οι Μαροκινοί. Έχουν πάρα πολλές ε, intelligence, πολλές πληροφορίες, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την πραγματικότητα στο Σαχέλ, είναι εντυπωσιακή η γνώση τους και τις μοιράζονται με τα κράτη, μέλη. Υπάρχει μια έντονη επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ του Μαρόκου, της Ισπανίας, της Γαλλίας και πολλών άλλων κρατών μελών. Και όπως ξέρετε το Μαρόκο θα είναι ε, το Δεκέμβριο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ε, θα είναι λοιπόν σημαντική η θέση του για την υιοθέτηση του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, που θα μας επιτρέψει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης. Το Μαρόκο είναι σημαντική δύναμη σε όλο το μηχανισμό και η Αλγερία βεβαίως είναι. Προηγουμένως σας μίλησα για την επιθυμία μας η Αλγερία να μπλοκάρει περισσότερο τη δυνατότητα ανεφοδιασμού των των τρομοκρατικών ομάδων μέσω αυξημένου ελέγχου των συνόρων. Ξέρετε πολύ καλά ότι ενεργοποιείται πολύ και στη διαμεσολάβηση. Είναι πολύ σημαντικός εταίρος και προσπαθούμε να κάνουμε πολλέ προσπάθειε πολλές προσπάθειες συντονισμού με την Αλγερία. για την επίπτωση του θανάτου του Μπιν Λάντεν. Ξέρετε πολύ καλά ότι το GSPC είχε τρομερές δυσκολίες στο παρελθόν. Έκανε μια προσπάθεια να, να αναδιοργανωθεί, να βρει νέους μαχητές και από το θάνατο του Μπιν Λάντεν όμως υπάρχει περιφερειοποίηση αυτής της ομάδας Δεν θα πρέπει όμως να πιστέψουμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει ο ίδιος συντονισμός σε επίπεδο της Αλκάιντα που υπήρχε παλιά. Αναλύσαμε αυτές τις περιφερειακές ομάδες, της Αλσάμπα, της ΑΚΜΗ, της αντίστοιχης ομάδας στην Ιεμένη, να, την, να, να τις καταλάβουμε με περιφερειακούς όρους. Ε, γιατί νομίζουμε ότι είναι πιο οργανωμένοι από ότι είναι. Ε, επίσης, πολλά από τα, τις προτεραιότητες είναι τοπικές των ομάδων αυτών. Ε, είναι όλο και πιο τοπική η εστίασή τους. Δεν, υπάρχει οδηγίες, δεν υπάρχουν οδηγίες ή άμεσα που περνάνε από το κέντρο στο ακμή. Από την άλλη όμως ε, η ομάδα αυτή απλώνεται σε όλη την Αφρική. Παρότι η αρχηγή της είναι Αλγερινή, απλώνεται στην υπόλοιπη Αφρική παράλληλα μετασχηματίζεται και τρομοκρατική δράση έχει και προσπαθεί ας πούμε να εξασφαλίσει και κοινωνικές υπηρεσίες στον πληθυσμό για να τους, για να τους ελέγξει. Επίσης αναπτύσσεται και στην αρχίζει να παίρνει και στοιχεία από, τους, από το ΦΑΡΚ της Κολομβίας. Επίσης, κρατημέλη κράτη-μέλη αρχίζουν να αναπτύσσουν συστήματα ασφαλείας στα αεροδρόμια γιατί φοβούνται πυράβλους μπορεί να τα πλήξουν τι κάνει η Υπηρεσία εξωτερική Δράσης για να εξασφαλίσει τις αποθήκες που υπάρχουν στη Λιβύη. Εγώ είχα επισημάνει τον κίνδυνο πριν από την κρίση της Λιβύης και ήθελα να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε και την ανάκτηση αλλά και την ασφάλεια των αποθηκών. Τώρα, για την διάδοση πυρηνικού υλικού, να προσθέσω σε αυτά που είπε ο συναδελφός μου ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης δημιουργεί αυτή τη στιγμή ένα κέντρο αριστείας. Κέντρα αριστείας σε όλο τον κόσμο. Ένα από τα οποία βρίσκεται στο Μαρόκο από ό,τι καταλαβαίνω. Το μέλος ο στόχος του είναι, ο στόχος του είναι να βοηθήσει τις χώρες περιοχής να δημιουργήσει τις απαραίτητες ε, πολιτικές για να αντιμετωπιστεί το σχάσιμο υλικό. Και το ουράνιο του Νίγηρα είναι πάρα πολύ σημαντικό από αυτή την άποψη και γι' αυτό το κέντρο αριστείας ελπίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ενεργό για τα θέματα αυτά. Για το ερώτημα του κυρίου ε, Κέλαμ νομίζω ότι απήντησα για την Αλγερία. Για τον προπολογισμό, αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό και ενδιαφέρον. Υπάρχει τώρα μια διαπραγμάτευση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τα εργαλεία χρηματοδότηση και ένα από του φόβου μου και ξέρω γιατί συζητά το θέμα αυτό και το κατανοώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, υπάρχει μια σκληρή συζήτηση για το ποσοστό που θα χρησιμοποιηθεί από το εργαλείο για την ε, σταθερότητα και τη χρήση των αναπτυξιακών πόρων. Λόγω της διαπραγμάτευσης φοβάμαι ότι οι φόροι, οι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα μειωθούν ιδιαίτερα. Στο τελευταίο μου έγγραφο συζήτησης που έστειλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μου, θέλω να εξηγήσω ότι πέραν της εντύπωσης που υπάρχει στις Βρυξέλλες ότι τα χρήματα ανάπτυξης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στόχους ασφαλείας μέσα στο πλαίσιο του ΩΣΑ, αυτό δεν ισχύει. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καθαρά συλλογή πληροφοριών από μυστικές υπηρεσίες, αλλά όλα τα άλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αναπτυξιακούς πόρους. Πιστεύω όμως ότι μέσα στα χρήματα που έχουμε για την ανάπτυξη θα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα κονδύλια για αντιτρομοκρατικές δράσεις. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θέλω να σας ε, επιστήσω την προσοχή. Μπορώ να σας δώσω διμερώς περισσότερες λεπτομέρειες γιατί κινδυνεύουμε να έχουμε λιγότερα χρήματα από το 2014 για αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ε, τέλος, εν τέλει, ο ουαχαμπισμός Πολύ καλό το ερώτημά σας και πολύ δύσκολο να το απαντήσω. Πρέπει να, να ασχοληθούμε περισσότερο με το θέμα αυτό. Εγώ θα είμαι στον πολιτικό διάλογο με τη Σαουδική Αραβία το Δεκέμβριο στα πλαίσια της ε, εγγενίασης του κέντρου αριστείας στο Αμπουντάμι. Αυτό να θέμα πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο. Η κυρία Γκόμες, χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο would rather ask... Ask uh, Manuel. Ο Μανουέλ μπορεί να πει περισσότερα. Ε, ε oui, oui, madame ε, κυρία Γκόμες, ήταν πολύ σημαντικό το ερώτημα αυτό. Και έχει να κάνει βέβαια και με τη γεωπολιτική και με τους περιφερειακούς οργανισμούς. Κατά κάποιο τρόπο, οι ηγέτες της Γουινέας Μπισάου, ο στρατός ουσιαστικά, οι οποίοι είναι κατά κάποιο τρόπο οι εμπειρογνώμονες marketing των καρτέλ ναρκωτικών, αυτοί βρίσκονται πάντα πίσω από οποιοδήποτε πραξικόπημα, πίσω από όλες τις φατρίες πολιτικών και στρατιωτικών, όλοι αυτοί είναι εμπεπλεγμένη στο εμπόριο ναρκωτικών. Αλλά ήταν πολύ αποτελεσματική στο να μπορέσουν να διχάσουν τους διάφορους περιφερειακούς οργανισμούς. Στην ε, Αγγόλα καταφέρανε να ε, αποκλείσουν την ΕΚΟΑ... την ε, Ένωση των Χωρών της Δυτικής Αφρικής από τη Γουινέα Μπισάου. Χωρίς αυτό τον φορέα λοιπόν, τον χρησιμοποίησαν στη συνέχεια εναντίον της Ένωσης των Κρατών της Περιοχής στην Αγγόλα. Σε επίπεδο λοιπόν διεθνούς κοινότητας εμείς είμαστε λίγο πίσω από την στροφή, πίσω από την καμπύλη. Δεν έχουμε προλάβει τα γεγονότα. Υπάρχει ο ανταγωνισμός της Νιγηρίας με την Αγγόλα και γι' αυτό έχουν πάρει μια στραβή θέση. Γιατί εμείς ε, δεν συμφωνούμε με την Ένωση των Κρατών της Δυτικής Αφρικής για τη Γουινέα Μπισάου, τη θέση που έχει αναλάβει. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και οι πέντε μας περιφερειακοί οργανισμοί, ο ΙΕ, η Αφρικανική Ένωση, η Ένωση της Δυτικής Αφρικής, η ΣΕΛΠ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να κάνουμε μια αποστολή εκεί πέρα. Αποστολή. Αλλά για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουμε μεταξύ μας για τους όρους αναφοράς, για μια κοινή ανάλυση και ένα κοινό στόχο. και επομένως τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουμε μια συνάντηση στην Αντισαμπέβα και μετά στην Αμπούτζα, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο οι πέντε αυτοί οι οργανισμοί θα έχουν κοινού όρους αναφοράς για αυτήν την αποστολή. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι η Ένωση των Κρατών της Δυτικής Αφρικής δεν πετυχαίνει αυτό που πρέπει να κάνει στη Γουινέα Μπισάου. Στο Μάλι είναι πιο αποτελεσματική, έχει βελτιωθεί η αντιμετώπιση της κρίσης και τους είπαμε ο, ο Επίτροπος Φλεϊμάν από την ECOWAS, από την Ένωση των Κρατών Αυτών της Ειδικής Αφρικής, τους εξηγήσαμε ποια είναι η ειδική μας ανάγνωση της κατάστασης στην, στην ε, Γουινέα Μπισάου και επειδή προέρχεται από την Ιγυρία η κυρία αυτή η επικεφαλής ήταν ε, είχε μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά τελικά ήταν πιο ανοιχτή και άκουσε και τα επιχείρηματά μας, τα επιχείρηματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τουλάχιστον ορισμένων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω λοιπόν ότι έτσι θα βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν ξέρω αν αυτό σας ικανοποιεί. Η κατάσταση δεν έχει ακόμα <clears throat> ξεδιαλυνθεί. Η μόνη λύση για τη Γουινέα Μπισάου είναι να υπάρξει μια εκαθάριση της στρατιωτικής ιεραρχίας εκεί και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με πολύ στεναρές δράσεις της διεθνούς κοινότητας. Μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γκέρνς πρωτού κλείσουμε. Ο κύριος Γκέρνς είναι ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας με τις χώρες της Δυτικής Αφρικής. Ήμουν πρόεδρος της ε, λέσχης του Σαχέλ, αλλά είναι περίπου ίδια γεωγραφική περιοχή. Θέλω να πω το εξή. στο τέλο τη παρέμβασή σα, κύριε Ντεκέρκοφ, μιλήσατε για τα ποσά τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν ε, ως αναπτυξιακή βοήθεια με βάση τους κανόνες τη Επιτροπής ε, του ΟΣΑ και κυρίως ε, εκείνα που δίδονται για τον τομέα της Άμυνα. Υπάρχει ένα προηγούμενο του 2002-2003, αν δεν απατώμε, όπου ευρωπαϊκά κονδύλια ανάπτυξης δόθηκαν στην Αφρικανική Ένωση Αυτά τα ποσά κανονικά ε, έπρεπε να είχαν πάει για να αναπτύξουν την, ε, ανάπ την διακυβέρνηση της Αφρικής. Δεν ήταν δηλαδή ποσά για επιχειρήσεις. Αν θυμάμαι καλά. Νομίζω όμως ότι αυτό το θέμα πρέπει να το συζητήσουμε ενδελεχώς. Δεν έχει νόημα να δίνουμε αναπτυξιακή βοήθεια για την άμυνα. Υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές που δεν πρέπει να υπερβαίνουμε, οι οποίες επιβάλλονται από τη σύνεση που πρέπει να υπάρχει ε, στην ανθρωπιστική βοήθεια. Συχνά λοιπόν ε, με αυτά τα κονδύλια ε, θεωρούμε ότι χρηματοδοτούμε ας πούμε ανθρωπιστικές οργανώσεις που βάζουν στρατιωτική στολή. Έτσι τους αντιλαμβάνονται οι πληθυσμοί. Πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα και θα πρέπει να βάλουμε κάποιες, κάποια σαφή όρια. Στο παρελθόν ήμουν υπεύθυνο και για θέματα άμυνας και για ανθρωπιστική βοήθεια βοήθεια για την ανάπτυξη, καταλαβαίνω τι ευαισθησίε και των μεν και των δε. Δεν είμαι μέλο τη Επιτροπή σα. δεν μπορούμε να είμαστε παντού σε όλε τι επιτροπέ, αλλά αν μπορώ να κάνω μια πρόταση, κύριε Ντανζόν, είναι να συζητήσετε λιγάκι αυτό το θέμα. Είμαι έτοιμο να συμμετάσχω στην, στον προβληματισμό όσο μπορώ. Να πω δύο λόγια γιατί πρέπει να γίνει μια προσπάθεια πέρα από την περιοχή που συζητάμε. Πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Κανονικά θα πρέπει να έχουμε πιο πολύ χρόνο. Θα προσπαθήσω να ετοιμάσω και ένα έγγραφο να και θα κοιτάξω όλα τα έγγραφα του ΩΣΑ, γιατί αυτά που ακούω να, λέγονται Βρυξέλη, να, ακούω, να λέγεται στις Βρυξέλλες είναι ότι αυτό δεν γίνεται, γιατί αντιτίθεται όσα αυτό δεν είναι αλήθεια. Ε, δεν υπάρχει πουθενά στα έγγραφα κάτι τέτοιο. Εμείς το λέμε προφορικά, αλλά τα έγγραφα δεν το λένε. Ε, φυσικά το νομικό επιχείρημα είναι ε, δεν είναι σωστό αυτό, δεν πρέπει να δοθούν λεφτά ανθρωπιστικής, αναπτυξιακής βοήθειας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εγώ δεν είπα... Και καταλαβαίνω τι λέτε για το ανθρωπιστικό θέμα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το ψάξουμε το θέμα, ειδικά στο, στο στη διαχείριση τη ασφάλεια, στον τομέα τη διαχείριση τη ασφάλεια. Εγώ και ο Μανουέλ ετοιμάσαμε μια στρατηγική για τη Σαχέλ και προσπαθούμε να έχουμε μια συνολική θεώρηση και να κινητοποιήσουμε όλα τα μέσα. Και ο Επίτροπο Πίμπαλκ χαίρομαι που συμφωνεί μαζί μα. 150 ε, εκατομμύρια ευρώ ε, επιπλέον για να υποστηρίξουμε τη στρατηγική της ΣΑΧΕΛ. Είμαστε σε καλό δρόμο. Καλό θα ήταν να γίνει αυτή η συζήτηση. Ε, Επίσης αυτό που είπατε, η ειρηνευτική συμφωνία για την Αφρική. Ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση, λέει ο Πρόεδρος. Θέλω να ευχαριστήσω τους τρεις ομιλητές μας για την ειλικρίνειά τους, για το ότι τα είπαν έξω από τα δόντια. Ε, αυτά που είπαν δεν ήταν πάντα έπαινοι προς τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν ήταν πραγματικά ειλικρινής. Έχω, μια... Έχω ένα πρόβλημα όμως. Έχω την αίσθηση ότι αυτά που κάνουμε που και λέμε τώρα θα πρέπει να τα είχαμε συζητήσει και κάνει πριν από τρία χρόνια. Να... Ε, θα πρέπει να είχαμε συζητήσει πώς ε, λειτουργούν κάποιες δομές. Νομίζω ότι έχουμε και τη γραφειοκρατία και την καθυστέρηση και την αναποφασιστικότητα που είχαμε και πιο παλιά. Καταλαβαίνω του λόγου που είπατε, τι εξηγήσει που είπατε. Ο κύριο Λόπε Μπλάνκο εξήγησε τι δυσκολίε για να δημιουργηθεί μια στρατηγική και η στρατηγική αυτή είναι αναγκαστικά συνοδευτική. Ε, συνοδεύει τι δράσει των τοπικών φορέων. Παρ' όλα αυτά, δεν θα έπρεπε, ε, εν τιαφή περιπτώσει αξίζει τον κόπο να έχουμε μια στρατηγική. Αν κάθε μέρα καταλαβαίνουμε και συνειδητοποιούμε ότι δεν έχουμε τα μέσα. Γιατί δημιουργούμε προσδοκίες, δυσανάλογες ε, στα μυαλά κάποιων και κυρίως ευρωβουλευτών. Και ακούμε να γίνεται λόγος για παγκόσμια προσέγγιση, για φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λέει και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος, για την προσθέμενη αξία που φέρνουμε εμείς σε αυτές τις περιοχές που χρειάζονται αυτή την παγκόσμια προσέγγιση, τη συνολική προσέγγιση ε, και συνειδητοποιούμε παράλληλα τα αντικειμενικά όρια των μέσων μας, των διαδικασιών μας. Το να λέμε το 2012 ότι έχουμε χρήματα, αλλά είναι δύσκολο να τα ξεμπλοκάρουμε αυτά τα χρήματα και να τα διοχετεύσουμε, δεν είναι πολύ σοβαρό σε σχέση με τις φιλοδοξίες που έχουμε πει ότι έχουμε εδώ και δύο χρόνια και με τις δομές που έχουν δημιουργηθεί στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Όλα αυτά δείχνουν κάποιε δυσκολίε, θα έλεγα. Αλλά για να το πω τόσο χοντρά, τέλο πάντων δυσκολίε που πρέπει να επιλύσουμε πολύ γρήγορα. Γιατί αν με αυτά τα, με αυτά τα παραδείγματα και με άλλα θέματα όπου χρειαζόμαστε να δράσουμε γρήγορα, αν δεν το κάνουμε, τότε η αξιοπιστία του όλου οικοδομήματος καταρακώνεται. Η συνθήκη είναι πολύ φιλόδοξη και μας δεσμεύει όλους. Τα κράτη-μέλη, καταρχήν, για θέματα επάνδρωσης και προσωπικού, επάνδρωσης των αποστολών ας πούμε, και των επιχειρήσεων, πρόβλημα που γίνεται όλο και πιο οξύ, αλλά είναι και πρόβλημα δομών. Ε, υπάρχει πρόβλημα με τις δομές της ΚΠΑ και δεν είναι φυσιολογικό το 2012 να μην είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και, δεν μπο, και να μην μπορούμε να αναπτύξουμε κάποιες ε, αποστολές που πρέπει να τις κάνουμε, αλλά που δεν είναι και γιγαντιές, εν Θα πρέπει να έχουμε τους επαρκείς πόρους για αυτές τις ε, αποστολές, στρατιωτικές και πολιτικές. Αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να την κάνουμε και να τη συνεχίσουμε την υπατή εκπρόσωπο, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Ευχαριστώ για την παρουσία σας πάντως, ευχαριστώ για την ειλικρίνειά σας, ευχαριστώ για τον προβληματισμό σας. Σας ευχαριστώ κυρίως εσάς, κύριε Λόπες Μπλάνκο, γιατί νομίζω ότι είναι η τελευταία φορά που έρχεστε σε αυτή την υποεπιτροπή, τουλάχιστον με αυτή την ιδιότητα. Ε, ίσως μετά την ε, σταξιοδότησή σας ε, που θα την πάρετε στο τέλος ε, του 2012 θα ξαναέρθετε ως εξωτερικός σύμβουλος να μας δώσετε τα φώτα σας για την Αφρική. Θα Σταματήσουμε τώρα τη συνεδρίασή μας για να συνεδριάσει το Προεδρείο και θα τα ξαναπούμε σήμερα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ όλους.